Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σα. Προτείνω να ξεκινήσουμε τι συνεδριάσει. Παρακαλώ, απόλυτη ησυχία να επικρατήσει την αίθουσα. Ευχαριστώ. Απόλυτη ησυχία, κυρία Συγκετρία. Παρακαλώ. Είδατε λοιπόν το σχέδιο, σχέδιο ημερησία για Εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσει λογίζεται ως βάση εργασία μας αυτό το σχέδιο ημερησίας διατάξεως. Και εγώ προτείνω από πλευρά μου δύο μικρές τροποποιήσεις, καταρχάς σε συνεργασία και συνεννόηση με τον εισηγητή κύριο Μπέγκε. Προτείνουμε να αναβληθούν τα σημεία 8 και 9 της ημερησίας διάταξης για την προσεχή μας συνεδρίαση. Πρόκειται για το περίφημο πακέτο Λισαβόνας που ονομαζόταν παλιά πακέτο Μπέγκε και πακέτο Λαμασούρ επίσης. Τώρα ονομάζεται πακέτο Λισαβόνα. Θα ξαναλλάξει φαντάζομαι όνομα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε αρκετά στοιχεία στη θέση μα για, να το χρησιμο... για να το συζητήσουμε ουσιαστικά και δεν έχουμε πάνω απ' όλα την γνωμοδότηση που έχουμε ζητήσει, την, γνωμάτευση μάλλον που έχουμε ζητήσει από την νομική μα υπηρεσία η οποία είναι άκρως απαραίτητη για να γίνει μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και στη συνέχεια να υιοθετηθεί η βασική μας θέση στα, και η θέση, η θέση επί τους, ε, καταρχήν θέση και η κατάρθρον θέση για την ε, σημαντική αυτή έκθεση. Επίσης η έκθεση How Can έχει, έχει επισημανθεί αυτό στην έκθεση στο Combo News και Αντιστρέφοντας τώρα τους όρους, και κερδίσουμε χρόνο μέχρι τα σημεία τη διάταξης, θα σας προτείνω η συζήτηση να ξεκινήσει από κοινού με τους δύο συνεισηγητές της Ταγματικής Επιτροπής ως προς την πρόταση τροποποίηση του άρθρου 136 της Συνθήκης, το σχετικό με τη λειτουργία της Ένωσης. Για τη συζήτηση αυτή έχουμε και καλωσορίζουμε παρόντες τον κύριο Έλμαν Μπρόκ, ε, συνεισηγητή από την Επιτροπή των Σταγματικών Υποθέσεων μαζί με τον συνάδελφο κύριο Γκουαλτιέρη, ο οποίος παραδόξως πως σήμερα φέρει το όνομα Κοτσολίνο στην κάρτα του. Αλλά είναι όπως το πακέτο της Λισαβόνας φαίνεται. Αλλάζει όνομα. Ο κύριος Κοτσολίνο λοιπόν. και ο κύριος Αλμαπλούκ. Αυτά προς την ημερήσια διάταξη. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, συγκρίνονται. Ανακοινώσεις. Στο πρώτο σημείο με στον ενθουσιασμό της ε, η Επιτροπή των Προϋπολογισμών έκρινε πως εγώ λόγω προσωπικών δεξιτήτων και ηλικία ήμουν ο καταλληλότερος για να διατυπώσω μια γραπτή επιστολή προς τον Πρόεδρο σχετική με το Ευρωπαϊκό Έτος για το Ενεργόν Γύρας το 2012 δηλαδή. Έγινε η επαλήθευση των τεχνικών στοιχείων, των πρακτικών στοιχείων από τη γραμματεία και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις θα υπογράψω την επιστολή της οποίας άλλωστε έχετε λάβει σχέδιο στους φακέλους σας για μια θετική γνωμοδότηση. Σχετική με το έτος 2012 και το ενεργόν γύρας. Εάν συμφωνείτε λοιπόν μπορούμε την επιστολή αυτή, αν υπάρχουν αντιρρήσει καλύτερα, να την υποβάλουμε σε ψηφοφορία. Υπάρχουν αντιρρήσει προ την επιστολή. Όχι. Καλώ λοιπόν. Επομένω θεωρούμε ότι εγκρίνεται η επιστολή και αναλαμβάνει ο Πρόεδρος να αποστείλει τη σχετική επιστολή εκ μέρους Επιτροπής των Προϋπολογισμών. Σας ευχαριστώ. Στις ανακοινώσεις. Έχετε επίσης λάβει, μάλλον έχουμε επίσης λάβει, και ίσως και εγώ, επιστολή του Πρόεδρου Μπούζεκ για την πρόοδο στην εφαρμογή του πιλωτικού σχεδίου 2011 Ευρωπαϊκή Στρατηγική και Πολιτική Ανάλυση. Ή καλύτερα σύστημα Ευρωπαϊκής Στρατηγικής και Πολιτικής Ανάλυσης. Πρόκειται για μια επιστολή άκουσα ενδιαφέρουσα, γιατί αποτελεί μια θετική και ανοιχτή ανταπόκριση από πλευρά του Πρόεδρου του Κοινοβουλίου σε μια πρωτοβουλία την οποία από κοινού προώθησαν τα τρία θεσμικά όργανα και αφού αποτέλεσε πιλωτικό σχέδιο για ένα πρώτο έτος, έχει σαν στόχο να μετατραπεί σε ένα μόνιμο όργανο και μόνιμη δραστηριότητα προς, στην υπηρεσία των τριών θεσμικών οργάνων. Θα ενθυμίστε ότι ο κύριος Σέμψελες ήταν ο πρώτος ο οποίος ανέλαβε αυτή την υπόθεση με ένα έγγραφο που κυκλοφορήσει. James Σέιλις διορθώνει η διερμηνέα. και θα πρότεινα ο κύριο Σέιλις να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις και τι, συνέχεια έχει αυτή η επιστολή. James. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ που περιλάβατε το θέμα αυτό στην ημερήσια τη Επιτροπή μας. Οφείλω να πω ότι ε, δημοσιονομικά είναι μάλλον ε, λόγος έκπληξης για μας ότι ένα τέτοιο θέμα εγγράφεται μέσα στον προπολογισμό. Ένα σύστημα λοιπόν για ένα διοργανικό σύστημα που θα υπολογίζει και θα καταγράφει μακροοικονομικές ε, τάσεις και ανάλυση των κύριων θεμάτων που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τα δημοσιονομικά θέματα. Αυτά λοιπόν σε συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής Συμβουλίου και Κοινοβουλίου και θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή για να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το σύστημα το 2012. Η επιστολή του Πρόεδρου Πούσεκ υπογραμμίζει νομίζω πολύ σύντομα τα εξή σημεία. Καταρχά τη διαδικασία, τη θέσπιση δηλαδή τη διαδικασία ε, τη Task Force με του ε, εισηγητέ τους εισηγητές και τη συνεργασία με, με την Υπηρεσία Εξωτερικών Σχέσεων. Επίση τη σύσταση κατευθυντηρίων γραμμών για την εφαρμογή των πιλωτικών προγραμμάτων και τη διάθεση των κονδυλίων που διατίθενται τώρα το 2011 και δεύτερον ο στόχος και η διαδικασία καλύτερα της EUISS αυτής, της, αυτού του οργάνου θα ήταν μέχρι το τέλος του 2011 ε, και μάλλον χάρη ε, με χρήση της διαδικασίας Λαμασούρ για να δημιουργηθεί ένα σύστημα, θα ετοιμάσει ένα έγγραφο σχετικό με την ανάλυση των δημοσιονομικών, οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών συνθήκων που αντιμετωπίζει το 2011 η Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης κύριες προκλήσεις και επιλογές που θα έχουν να αντιμετωπίσουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στον επόμενο διοργανικό κύκλο 2014 έως 2019. Άρα ο μακροπρόθεσμος στόχος αυτού του πιλωτικού σχεδίου είναι να αναπτυχθεί η συνήθεια, το ήθος δηλαδή της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων, ώστε και η Ευρωπαϊκή Ένωση να ωφεληθεί από καλύτερη ανάλυση, συνεργασία, επιλογές μεταξύ των διαφόρων προκλήσεων και εναλλακτικών. Και με κύρια ιδέα ε, αυτό το σύστημα να, να αναφέρεται ως Ευρωπαϊκό Σύστημα Στρατηγικής και Πολιτικής Ανάλυσης. Και για να ολοκληρώνω, ε, εάν αναστευτεί με επιτυχία αυτό το σχέδιο, θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δυνάμει του άρθρου 49, αν δεν απατώμε, να προτείνει την θεσμοθέτησή του σε μια πιο μόνιμη δομή. Αυτό ανάλογα με το πώς θα προχωρήσει και θα εξελιχθεί το σχέδιο. Επίσης, Έχω καλέσει και τα αρμόδια θεσμικά όργανα να συμμετάσχουν στη διαδικασία αυτή. Αν δεν έχει αντίρρηση η Επιτροπή των Προπολογισμών, θα συνεχίσω αυτή τη ε, συνεργασία και νομίζω ότι ήρθε η ώρα πια η Επιτροπή μα να έχει μια πιο ε, στοχευμένη και στρατηγική εξέταση στην υπόθεση αυτή και όχι μόνο περιστασιακή. Ευχαριστώ πολύ, Τζέιμ. Ε, εξαιρετική αυτή η εργασία σας όπως ε, υπενθύμησες βεβαίως εξαρτηθεί πρώτα από τον τρόπο με τον οποίο το πιλωτικό πρόγραμμα θα εκτελεστεί. Έχουμε όμως κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η φάση καθίδρυσης ε, της νέας διαδικασίας του νέου οργάνου και είναι πάρα πολύ σημαντική η διαδικασία για τα τρία θεσμικά όργανα να ε, μάθουμε να εργαζόμαστε με μια μακροχρόνια διάσταση και προοπτική. Έχουν επίγνωση αυτού και τα τρία θεσμικά όρα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Γενικός Γραμματέας παρακολουθούν ε, και για τον επόμενο προϋπολογισμό και ο Τζέιμς σε στενή συνεργασία με την εισηγήτρια του 2000 12 τη Φραντσέσκα, καθώς επίσης και τον εισηγητή τη Επιτροπής Σούρε που δεν έχει φτάσει ακόμα για την ε, βιώσιμη και φορο χρηματοδότηση. Υπόλοιπε ανακοινώσεις του Προέδρου εντάχει. Έχετε το κόμπο με τις γλώσσες και στο διαδίκτυο απευθείας επίσης. Βλέπετε τους συνδέσμους ε, για το που θα βρείτε για την εκτέλεση του προπολογισμού 2010 τα έγγραφα στο διαδίκτυο και έρχομαι στο σημείο... Α, συγγνώμη, διακόπτει ο πρόεδρος. Πρέπει επίσης να σας πω ότι λάβαμε και σας έχω διαβιβάσει από 3 Φεβρουαρίου μια επιστολή, αντίγραφο δηλαδή, της επιστολής του Επιτρόπου Λεβαντόφσκι προς όλους τους προέδρους όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων συμπεριλαμβανομένου λοιπόν και του Προέδρου Μπούζεκ, όπου εκφράζει την αίσθησή του και ευγενικά κάνει κάποιες συστάσεις ως Πρόεδρος των Θεσμικών Οργάνων για να προετοιμάσουν αντίστοιχα το προσχέδιο του λειτουργικού του προπολογισμού για το 2012, του κάθε θεσμικό όργανο. Θυμίζοντας ότι είναι πάρα πολύ σφιχτά τα οικονομικά μας, και όλα τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να περιορίσουν ε, τις λειτουργικές τους δαπάνες. Έχει και τη φιλοδοξία να δώσει το παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επιθυμεί αντιστοίχως να πράξουν και τα άλλα θεσμικά όργανα με ισορροπία. Σημείο 3 έγκριση των πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων. Ε, γρήγορα θα το διεκπαιρεώσουμε διότι πρακτικά δεν έχουμε. Και περνούμε στο σημείο 3α, δηλαδή παρουσίες εκ μέρους των συνεισηγητών της ε, Συνταγματικής Επιτροπής της πρώτας τροποποίησης της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μεγαλύτερη δημοσιονομική πειθαρχία και τη νέα διαδικασία του λεγόμενου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Δύο είναι οι συγητές, συν ο κύριο Γκουαλτιέρη, παρακαλώ, πρώτο και μετά ο κύριο Μπροκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Από κοινού με τον συνάδελφο Μπροκ κρίναμε σκόπιμο να ζητήσουμε να σας παρουσιάσουμε το θέμα αυτό στην Επιτροπή σας. Διότι θεωρούμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει πολλές πλευρές και εμπολής αφορά και την Επιτροπή σας. Ξέρετε ότι με βάση την απλοποιημένη διαδικασία της αναθεωρημένης συνθήκης 4806 το Κοινοβούλιο πρέπει να γνωμοδοτήσει σχετικά με την μεταρρύθμιση που το Συμβούλιο την προτάσει του Βελγίου ήδη συμφώνησε στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου για αναθεώρηση του άρθρου 136 της συνθήκης. Αυτή η, πρώτη η πρόταση αναθεώρησης απαιτεί τα κράτη-μέλη που έχουν το ευρώ να μπορούν να έχουν ένα μηχανισμό οι ημερομηνίε κλπ. υπό ορισμένου όρους χώρες σε σχέση με το ευρώ. Θεωρήσουμε χρήσιμη μια ανταλλαγή απόψεων. Αν και η Επιτροπή Προπολογισμών δεν είναι η κύρια επιτροπή, γιατί εμείς στην ΑΦΚΟ είμαστε η κύρια επιτροπή και υπάρχει γνωμοδότηση και της ε, Οικονομικής Επιτροπής. Αλλά το θέμα αυτό είναι κομβικό για γενικότερες και ευρύτερε συζητήσει που γίνονται αυτές τις μέρες για την οικονομική διακυβέρνηση της Ένωσης και γενικότερα για το μέλλον της Ένωσης. Φυσικά, εμείς θα φροντίσουμε να κινηθούμε με απόλυτο πνεύμα ευθύνης, επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ λεπτό. Ευθύνη βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν θα φροντίσουμε να εκπληρωθεί η υποχρέωση του Κοινοβουλίου να αναλύσει, να συζητήσει τα προβλήματα μια τόσο σημαντικής διαδικασίας όπως η αναθεώρηση της συνθήκης Λισαβόνας. Για τα διαδικαστικά προβλήματα δεν θα πω τίποτα. Ούτε για τις πολιτικές επιπτώσεις μιας διαδικασίας που απαιτεί 27 επικυρώσεις από 27 χώρες που μπορεί να κρατάνε την Ένωση με κομμένη την Ανάσα μέχρι το 2013 και τα Εθνικά Κοινοβούλια κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσαν να μπουν στη θέση του να ξαναρχίσουν να διαπραγματεύσει, να μπορούν να εκβιάσουν την Ένωση. Γιατί αν σταματήσει η διαδικασία επικύρωση, αυτό θα είχε καταστροφικέ συνέπειε, Οντολογικού χαρακτήρα θα έλεγα, υπαρξιακού μάλλον χαρακτήρα για την ίδια την Ένωση. Αυτέ είναι συνταγματικέ παρατηρήσει. Εμεί όμω, περισσότερο θέλουμε να σα παρουσιάσουμε ένα άλλο θέμα θέμα ουσίας. Συζητήθηκαν όλα αυτά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η συγκεκριμένη πρόταση περιγράφει έναν εντελά, εντελώς καθαρά διακυβερνητικό μηχανισμό, έξω δηλαδή από τις δομές της Ένωσης. Ο Αυτός ο μηχανισμός που κινήθηκε με διαφορετική ε, νομική βάση, το 122.2 της συνθήκης. προηγούμενη διαδικασία ήταν πρώτες της Κομισιόν, κοινοτική διαδικασία, 60 δις που τεγκιάται ο Ευρωπαϊκός Περιπολογισμός. Με τη μεταρρύθμιση όμως της συνθήκης, αυτός ο ισχύων μηχανισμός θα κηρυχθεί αντισυνταγματικός, θα απαγορευτεί η χρήση του. Μέχρι ότου βέβαια να ισχύσει ο επόμενος κανονισμός. Οπότε, ο ισχύων μηχανισμός που ξεκίνησε τον περασμένο Μάιο θα αντικατασταθεί από ένα μηχανισμό που τον δημιουργούν αποκλειστικά τα κράτη-μέλη μεταξύ τους, έξω από τον θεσμικό συνταγματικό ιστό της Ένωσης και έξω από την κοινωτική μέθοδο, όπως λέμε. αυτό για το Ευρωκοινοβούλιο θέτει προβλήματα. Είδαμε στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μια πρόταση για το σύμφωνο ανταγωνιστικότητας. Μπορεί να υπάρχουν πολλές απόψεις πάνω στο θέμα αυτό, έχει όμως το χαρακτηριστικό ότι και αυτό, τουλάχιστον το πρώτο αυτό σχέδιο πρότασης, σε διακυβερνητικό επίπεδο. Αυτή λοιπόν η τάση από τη μια μεριά θετική να ενισχύεται η οικονομική διακυβέρνηση, από την άλλη όμως να δημιουργούνται μορφώματα έξω από τον κοινωνικό ιστό, δημιουργεί προβλήματα και υποχρεώσεις. Σε σχέση με το ρόλο και την επίπτωση του κοινωνικού προπολογισμού, τη σχέση πρέπει να έχει ο προπολογισμό με διαδικασίε οικονομική διακυβέρνηση και στη σχέση ανάμεσα στη διαπραγμάτευση για το επόμενο MFF και τις διαδικασίες επικύρωσης με προθεσμία και τον 2 το 2013. Πολλοί συσχετισμοί λοιπόν, σχέσεις μάλλον, οι οποίε θα πρέπει να μας κάνουν στο Ευρωκοινοβούλιο να προβληματιστούμε. Τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτού του είδους η μεταρρύθμιση. Ακόμα δεν έχουμε κάνει σχέδιο εμείς. Εμείς ήρθαμε για να ακούσουμε σήμερα. Η πρόθεσή μας είναι να φροντίσουμε να ενισχυθεί η κοινωτική μέθοδος από τη μια μεριά και από την άλλη να είμαστε υπεύθυνοι σε ένα σημαντικό πέρασμα που είναι σημαντικό για τη σταθερότητα και το μέλλον του ευρώ. Πρόεδρος. Ε, Ευχαριστώ, αγαπητέ συνάδελφο ε, Μπρόκ. Ε, κύριε Πρόεδρε, μερικές συμπληρωματικές αν μου επιτρέπετε. Γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε εδώ ενώπιον μιας κατάστασης που συνδέεται με πολλούς ε, έτσι, αναγκαστικούς χειρισμούς και δεν χαρακτηρίζεται πάρα πολύ από νυφάλες και αντικειμενικές στάσεις. Κάποιο κράτος θεωρεί ότι χρειάζεται αλλαγή το πρωτογενές δίκαιο. Γιατί δεν μπορεί λόγω της ρήτρας bailout το συνταγματικό της δικαστήριο να ε, καταργήσει την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ναι, δεν ακούγεται ο κύριος Μπρόκ, το μικρόφωνο του είναι μακριά. Μάλιστα. Επαναλαμβάνω. Έχουμε λοιπόν κάποιες ε, καταστάσεις που μας αναγκάζουν να προχωρήσουμε με τρόπο λίγο αντικειμενικό και νυφάλιο. Γιατί σε ένα κράτος μέλος, που το γνωρίζω καλύτερα από τα υπόλοιπα, ε, ε, κυκλοφορεί και επικρατεί η άποψη ότι πρέπει να αλλάξει το πρωτογενές δίκαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. για να μην μπορεί το δικαστήριο, λόγω, ε, το συνταγματικό της χώρας, λόγω της Ρίτας Μπέιλαουλ να καταργεί το ευρωπαϊκό δίκαιο ε, ε, με αποφάσεις ομπρέλα κάθε φορά. Και αυτό έχει και πολιτικές επιπτώσεις. Δεύτερο, για να ασφαλιστεί, να εξασφαλιστεί το ευρώ, λένε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας μηχανισμός προστασίας, ομπρέλα, όποιος και να είναι αυτός, και μάλιστα ομόφωνα. Ένα τρίτο τώρα αυτό συνδέεται με μια σχετική ασφάλεια, παρόλα τα προβλήματα που ανέφερε ο Ροπέρτο, μόνο με μια απλουστευμένη διαδικασία. Γιατί αν ήταν αυτή η συνήθις κανονική διαδικασία να αναθεώρησης θήκη με συνταγματική, συντακτική συνέλευση κτλ. Θα ήταν κάτι απαγορευτικό για μας λόγω των καταστάσεων που επικρατούν στις αγορές. Τι σημαίνουν αυτά τώρα ξανά. Αυτό τι σημαίνει. Κάτι που και πάλι δεν καταλαβαίνω. Λιγότερο δηλαδή από τα προηγούμενα. Δηλαδή, οποιαδήποτε αλλαγή στις εξουσίες και στις αρμοδιότητες αυτόματα θα πρέπει να οδηγούν σε δημοψήφισμα, λέει μια άλλη χώρα. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατό να προσθεθεί η εξής πρόταση στη συνθήκη. όχι στην παράγραφο 1 του 136, γιατί αυτό θα σήμαινε, λέει, ενίσχυση των εξουσιών του Συμβουλίου. Και ανταυτού θα πρέπει να μπει σε ένα νέο εδάφιο, υπαριθμών 3, όπου γίνεται λόγος μόνο για τα κράτη-μέλη και όχι για το Συμβούλιο. Εξ όλων αυτών τώρα προκύπτει εξή κατάσταση που θα πρέπει να μας προβληματίσει. Πώς προχωρεί η διακυβερνητική ε, συνεργασία ε, σε τέτοιο βαθμό που δεν συνδέεται καν με τις κοινωνικές διαδικασίες. Γιατί στο παρελθόν στις διακυβερνητικές λύσεις ε, από κοινού ε, τα κράτη ανέθεταν σε ένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο να ε, κάνει τις αλλαγές αυτές, δεν ξέρω να τις παρακολουθήσει, να τις συνοδεύει, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό. Και αυτή τη στιγμή είχαν λυθεί όλα αυτά ε, σταδιακά να μπουν, να κατοχυρωθούν στη συνθήκη και να εφαρμόζονται ως κοινοτική πολιτική. Εάν τώρα είναι η πρόθεση συνειδητά να γίνουν όλα αυτά εκτός και ερήμην των θεσμικών οργάνων, υπάρχει ο εξή κίνδυνος. μπορούν να αναπτυχθούν τελείως νέες θεσμικές ε, δυνάμει και οντότητε που να μην έχουν σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πάλι κυκλοφορεί ένα όραμα που προέρχεται από τη χώρα που γνωρίζω καλύτερα εγώ για την πρόταση για το σύμφωνο ανταγωνιστικότητα. Δεν γίνεται καθόλου λόγος πλέον για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι θα πρέπει ε, μάλλον θα επιτρέπεται να κάνει ανάλυση μετά από 12 μήνες και να συγκαλέσει συνέλευση ε, των Εθνικών Κοινοβουλίων για παρακολούθηση των οικονομικών θεμάτων. Αν αυτά ε, γινόντουσαν πραγματικότητα, υπό την πίεση των αναγκών των αγορών, θα είχαμε και νέα εξέλιξη και νέα έτσι, καταναγκαστική εξέλιξη που με ανισχύει πάρα πολύ. Και αν το συνδέσω και με άλλα θέματα που έχουν άμεση ή έμεση σχέση και με τους νέους πόρους του προπολογισμού που τα έχουμε συζητήσει, τότε καταλαβαίνουμε πού βρισκόμαστε. Πώς έχει η κατάσταση. Ε, βέβαια δεν μπορούμε να το συζητάμε και στο Δινικές 24 και 25 Μαρτίου συνεδριάζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και αν δεν αποφασίσει γιατί δεν μπορεί να αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση εγώ δεν θέλω να ζήσω στις 27 ε, Μαρτίου τις αγορές ε, τι σημαίνει αυτό η μόνη προθεσμία για την γνωμοδότησή μας μάλλον αυτή η προθεσμία είναι η μόνη δυνατότητα που έχουμε να ασκήσουμε πίεση δεν ξέρω αν έχουμε το περιθώριο και την πολυτέλεια για λόγους ευθύνη να χάσουμε αυτή την προθεσμία τη 24 η 25 Αυτός είναι ο χρονικός στενός κορσές που έχουμε. Αλλά η ευθύνη δεν θα πρέπει να είναι μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και στα κρατημέλη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για το λόγο αυτό, παρακαλώ να καθίσουμε όλοι να σκεφτούμε το εξής. Με ποιο τρόπο μπορούμε στο πλαίσιο αυτό να εργαστούμε, να προβληματιστούμε και Βέβαια, καταλαβαίνω έτσι όπως έχουν οι καταστάσεις τώρα, δεν μπορούμε να αποφύγουμε τελείως τη διακυβερνητική συνεργασία, αλλά να δημιουργήσουμε γέφυρες και προς τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και προς την κοινοτική μέθοδο, να τα παρακολουθούμε, να τα συνοδεύουμε, να τα πλαισιώνουμε όπως και στο παρελθόν και θα παρακαλούσα τη γνώμη σας. Έκανε κάποιες προτάσεις ο Ρομπέρτο θα μπορούσα να τις υποστηρίξω. Και εγώ θα προτιμούσα την παράγραφο 1 και τις ρήτρες ευελιξίας και θεωρώ ότι και η ενισχυμένη συνεργασία θα μπορούσε να παίξει μεγαλύτερο ρόλο τα θεσμικά όργανα, αλλά πρέπει να σας πω για τους λόγους που προανέφερα, θεωρώ ότι είναι αρκετά περιορισμένο το περιθώριο ελιγμών, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές και παρακαλώ να το σκεφτούμε αυτό. Και κατά πόσο έχουμε κοινή άποψη στο Κοινοβούλιο και η δική μας Επιτροπή να κάνουμε και τις συζητήσεις τις επόμενες εβδομάδες έτσι με κάποιο κύρος και με κάποια ευθύνη. Κατά τα άλλα, έχουμε και την πρόθεση να χρησιμοποιήσουμε και την έκθεση και το αντίστοιχο ψήφισμα ε, για να ε, ακολουθήσουμε και το συνολικό πακέτο για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, για το Σύμφωνο ε, Ανταγωνιστικότητας, για τους ιδίους πόρους κτλ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει μια συνολική θεώρηση για όλα αυτά τα θέματα με ψήφισμα και αυτό χρειάζομαι και χρειαζόμαστε και την εμπειρία και τη γνώση της Επιτροπής αυτής. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Κάποιοι συνάδελφοι έχουν στήσει το λόγο ήδη. Για μόνο διευκρίνηση ως προς το χρονοδιάγραμμα για να δούμε ποιο χρονοδιάγραμμα προβλέπετε για την έγκριση επιδοσταγματικής επιτροπής αφενός και έγκριση και του ψηφίσματος αλλά και της γνωμοδότησης Ταγματικής Επιτροπής ε, για την αναθεώρηση της συνθήκης και νομοθετικού σχεδίου που σχετίζεται με το όλο σύνολο μέτρων. Παρακαλώ, κύριε Γκουαλτιέρη. Όπως μας θύμισε ο συνάδελφος Μπροκ, το Συμβούλιο μας ζητάει να το επιτρέψουμε να προχωρήσει στην έγκριση της τροποποίησης της συνθήκης στη συνεδρίαση 24 και 25 Μαρτίου. Αρχικά σήμαινε πολύ στριμωγμένο χρονοδιάγραμμα, γνωμοδέτηση του Κοινοβουλίου στην Ολομέλεια την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου και μετά η διαδικασία που θα ακολουθούσε. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τον Μάρτιο 1 ως υπόθεση εργασίας. Φροντίζοντας να εξασφαλιστεί ευρεία συζήτηση στο Κοινοβούλιο και με τα άλλα θεσμικά όργανα που θα πρέπει και αυτά να γνωμοδοτήσουν. ως ε, δεύτερη θέση, αν δεν το πετύχουμε αυτό, θα μπορούσαμε να είχαμε μια έγκριση στην ε, σύντομη σύνοδο, Μάρτιος 2. Και αμέσως μετά είναι το Συμβούλιο 24 του μηνός. Αυτά για το δικό μας χρονοδιάγραμμα. Τώρα για τις έξι προτάσεις. Ο πρόεδρος Μπούζεκ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεσμεύτηκε για μια γρήγορη διαδικασία. Δεν είμαι ε, εμπειρογνώμονας, αλλά νομίζω ότι έχουμε περισσότερο χρόνο εδώ. Και εδώ δεν έχουμε τον Μάρτιο ως καταληκτικό μήνα. Για την Επιτροπή ΑΦΚΟ και εικόν. τι θα μας πείτε. Κοιτάξτε, η ΕΚΟΝ ήδη ξεπέρασε, πέρασε την διαδικασία, την ε, ημερομηνία για, τους, ε, για τις ε, τροπολογίες. Είμαστε στις συμβατικές τροπολογίες. Δεν ξέρω πότε θα γίνει η ψήφιση. Αυτά για την ΕΚΟΝ, η οικονομική για την ΑΦΚΟ, Συνταγματική Επιτροπή. Έχουμε μία συνεδρίαση στις 14 του μηνός, όπου θα συζητηθεί το σχέδιο που θα παρουσιάσουμε. Η ψηφοφορία στην Συνταγματική Επιτροπή ή σε έκτακτη σύνοδο στο Στρασβούργο 1 τη Δευτέρα για ψήφο την Πέμπτη ή την επόμενη εβδομάδα των Επιτροπών 14-17. Οπότε θα ψηφίσουμε στην μικρή Ολομέλεια του Μαρτίου 2. Πολύ καλά. Θεωρητικά όλα αυτά και για λόγους που ανάφερε ο κύριος Μπρόκ πρέπει οπωσδήποτε να κινηθούμε αυτό το πνεύμα. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ τον ε, εισηγητή. Ο κύριος Άλβαρο έχει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Και ευχαριστώ τους συναδέλφους Γκουαλτιέρη και κυρίως τον κύριο Μπρόκ για την άκρος ενδιαφέρουσα ανάλυση. Και ιδιαίτερα για κύριο το κράτο μέλος που γνωρίζουμε καλύτερο κύριο κύριος Μπρόκ και εγώ. Έτσι είναι πιο εύκολα τα πράγματα, τα καταλαβαίνουμε πιο καλά. Θα ήθελα λοιπόν να δω πώς σκοπεύει το Συμβούλιο να αξιολογήσει αυτήν την κατάσταση και τις δυνάμεις του πάνω απ' όλα. Γιατί έχουμε τις προθεσμίες, αν κατάλαβα καλά το Κοινοβούλιο, εάν δεν γνωμοδοτεί στο Κοινοβούλιο το Συμβούλιο, μένει με δεμένα τα χέρια, άρα κατά κάποιο τρόπο εξαρτάται από το Κοινοβούλιο και άρα έχουμε κάθε συμφέρον και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ιδιαίτερα στο θέμα της περαιτέρω ε, οικονομικής ε, στονιστικής προσπάθειας, του οικονομικού στονισμού δηλαδή και κυρίως το θέμα της ε, ανταγωνιστικότητας, να εξασφαλίσουμε λύσεις οι οποίες και με διακυβερνητικό τρόπο θα μπορέσουν να λειτουργήσουν και σε συνεργασία με τα τυρά κοινοβουλία από τους που θα λειτουργούν. Και ίσως θα ήταν λύση το να γίνει η τροποποίηση του προτάσεως του Συμβουλίου μέσα από ε, ένα κείμενο, μια φράση που θα εισαγάγαμε στο δικό μας ψήφισμα. Έχει γίνει στο παρελθόν, υπάρχει προηγούμενο και ως εκ τούτου στο θέμα της ανταγωνιστικότητας, συμφώνου σταθερότητας η συμμετοχή του Κοινοβουλίου θα μπορούσε να συμπεριληφθεί ε, σαν στόχος για το Συμβούλιο ή σαν ε, παραδεδεγμένο στόχος του, του Συμβουλίου καλύτερα, ε, και να μπει έτσι μέσα στο δικό μας κείμενο και με αυτόν τον τρόπο να τροποποιηθεί η πρόταση του Συμβουλίου. Και έτσι θα είναι απόλυτα εφικτή. Επίσης θα πρέπει να δούμε αν πρόκειται να εισαχθούν ε, συστήματα κυρώσεων σε συνάρτηση με το άρθρο 136, αν αυτά θα λειτουργούν κατά τρόπο αυτοματοποιημένο, εάν δηλαδή αυτέ οι ποινέ θα τίθενται σε ισχύ αυτομάτω, εάν θα πρέπει να παρέμβει το Συμβούλιο. Ο πρόεδρο. ευχαριστώ. Η κυρία Τρίπελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τους δύο εμπειρογνώμονές μας, συναδέλφους. Θα ήθελα και εγώ να σταθώ στο ερώτημα που έθεσε ο κύριος Άλβαρο. Αν κατάλαβα καλά τα όσα άκουσα, καθοριστική σημασία σύνοδος για το θέμα του οικονομικού πακέτου, συμφωνού ανταγωνιστικότητας, είναι αυτή η σύνοδος της 23-24 Μαρτίου και χρειάζεται η στάση του Κοινοβουλίου να είναι τέτοια ώστε να πιέσουμε να μην επικρατήσει η τάση για διακυβερνητική συνεργασία που βάζει στο περιθώριο το Κοινοβούλιο, γιατί ό,τι δεν μπορεί να είναι προ το συμφέρον μα. Αυτό που προτείνει λοιπόν ο κύριο Άλβαρο θα ήταν μια λύση, αν έχουμε έναν τρόπο να προσδιορίσουμε εμεί συνθήκε υπό τι οποίε θα γίνει αυτό, τηρώντα τι προθεσμίε που έχουμε ε, να τηρήσουμε εφόσον επομιστήκαμε τη σύνταξη του κειμένου και Ίσως θα μπορούσαμε πολύ ξεκάθαρα για να μην ξεπέσουμε σε φιλολογίες και θεωρητικές ε, τοποθετήσεις, να διατυπώσουμε ένα κείμενο το οποίο πράγματι να είναι χρήσιμο και εποφελές για τις δύο πλευρές, ένα deal θα λέγαμε, έτσι ώστε και εμείς να διαφυλάξουμε τη θέση μας στις διαδικασίες αυτές και στην πολιτική αξιολόγηση ε, των ε, περιθωρίων που υπάρχουν, αλλά και ως προς την αξιολόγηση των ε, δεδομένων και των συγκεκριμένων διατυπώσεων. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο Κάλφιν. Πρόεδρε, το πρόβλημα δεν έγκυται μόνο στις τροπολογίες ή στον τρόπο αναθεώρησης συνθήκης Λισαβόνας, αλλά και στις αρμοδιότητες που εξέτασε το τελευταίο συμβούλιο. Εγώ προσωπικώς είμαι επιφυλακτικός, γιατί θεωρώ ότι μια τέτοια τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στην οικονομική σταθερότητα, ούτε καν στη ζώνη του ευρώ. Αυτή τη στιγμή έχουμε διακυβερνητικό συντονισμό. Το Συμβούλιο δηλαδή προτείνει τώρα έναν συντονισμό πιο έντονο, που όμως δεν αρκεί πάλι, δεν θα έχει επαρκή απήχηση ή επαρκή αντίκτυπο. Πιστεύω όμως ότι θα μπορούσαμε να επιμείνουμε και να πιέσουμε για μια λύση και για τη ζώνη του ευρώ, ε, πιο γενική, μια λύση πιο περιεκτική που να καλύπτει όχι μόνο τα κράτη της ζώνης του ευρώ αλλά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι να χαρακτηρίζει την πολιτική της κοινότητας εν γέννη. Ευχαριστώ που επιτρέπετε τη συζήτηση αυτή στο θέμα στην Επιτροπή των Προπολογισμών, γιατί και το, και το Συμβούλιο και η Επιτροπή εμένουν στην ιδέα ότι το μέσο αυτό στήριξης ε, αποτελεί αντίβαρος προς τον προϋπολογισμό. Αλλά αυτό δεν μπορεί να συμβεί παρά μόνο εάν ο προπολογισμό εξασφαλίζει τι απαραίτητε εγγυήσει για τη λειτουργία του συστήματο. Και ω εκ τούτου κάθε όφελος έχουμε όλοι και από τη διαφύλαξη τη δημοσιονομική σταθερότητα και της ε, άμεμπτης λειτουργίας του προπολογισμού και η ασδήποτε πρόταση αντιβαίνει αυτή την ε, αρχή της σταθερότητας γιατί η Φερρυπίν ενισχύει τον, τους κινδύνους ή περιορίζει μέσα. Επίσης, εάν τα θεσμικά όργανα δεν συμμετέχουν στην επίλυση των μεγάλων προβλημάτων, αυτομάτως ε, ε, πλήττεται το κύρος ε, και η αξιοπιστία τους και ως εκ τούτου θα πρέπει να αναλάβουμε δράση με βάση τους μηχανισμούς που έχουμε στη θέση μας ήδη. Ο κύριος Σούριαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι το θέμα της σταθερότητας του ευρώ συνδέεται πολύ στενά με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Επιτρέψτε μου να επανέλθω σε αυτό το ζήτημα και τώρα και στη συνέχεια συνεδρίαση των συντονιστών. Το Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να είναι μέρος του προβλήματος, αλλά μέρος της λύσης. Θα πρέπει να βοηθήσουμε στην εξέβρεση λύσης, γιατί πολύ εύκολα μπορεί να δημιουργηθεί εντύπωση ότι οι κυβερνήσεις προσπαθούν να βρουν μια λύση έτσι, διακυβερνητική, αντί να αναζητήσουν διοργανική λύση μέσα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Συμφωνώ με αυτό που υπόθηκε. Δεν θα ήταν καλή μια τέτοια λύση. Ούτε δημοκρατική. Θέλω και εγώ να λυθεί διαφορετικά το πρόβλημα. Και όπως ακούσαμε υπάρχει και εναλλακτική πρόταση να μην ε, οδηγήσουμε τη διαδικασία σε εμπλοκή, να μην παρεμποδίσουμε τα πράγματα και εν ώψη της Συνόδου του Μαρτιού, όπως είπε και ο Έλμαρ Μπροκ. Και η Χέλγα Τρούπελ. είναι υπέρ της ευρωπαϊκής σταθερότητας. Συμφωνώ απολύτως, λέει κυρία ε, κύριε Πρόεδρε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και στρατηγική σημασία. Ακούσαμε όλη αυτή τη συζήτηση για τον προπολογισμό και των ιδίων πόρων, ότι θα υπάρξει διαβούλευση του Κοινοβουλίου με άλλη μορφή όμως με άλλο τρόπο από εκείνο που εμείς επιθυμούσαμε, δηλαδή να έχουμε πλήρη συμμετοχή. Για το θέμα αυτό όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να ασκήσουμε την απαραίτητη πίεση για να μην μας παρακάμψουν. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα θεωρώ και εγώ ότι δεν πρέπει να χάσουμε καθόλου χρόνο. 24 Μαρτίου πάρα πολύ αργά. Ας προσπαθήσουμε να εγκρίνουμε στην πρώτη σύνοδο του Μαρτίου ε, την απόφαση αυτή και να αξιοποιήσουμε το διάστημα μέχρι τότε ε, για να χαράξουμε μια στρατηγική σημαίνουσα γιατί αυτό είναι και προς όφελος της σταθερότητας του ευρώ. Αν δεν είμαστε σε θέση εκεί να κάνουμε τη φωνή του Κοινοβουλίου να ακουστεί, θα είναι εξίσου σοβαρό με την υπόθεση SWIFT, όπως είπε ο κύριος Άλβαρο, ή ε, τα άλλα που αναγκαστήκαμε να κάνουμε τις για τον προϋπολογισμό. Πάντως θα πρέπει να έχει βαρύνουσα άποψη και θέση στο Κοινοβούλιο και να χαράξουμε τέτοια στρατηγική. Ευχαριστώ Ιζαπέλ. Ο κύριος Μπόκρος. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα. Δεν νομίζω ότι το, αυτή η ιδέα περί ανταγωνιστικότητας δεν πρέπει να το δούμε αν δίνει περισσότερες ή λιγότερες εξουσίες στο Κοινοβούλιο. Επίσης, δεν πιστεύω ότι δεν πρέπει να τη δούμε και από την σκοπιά του προπολογισμού. Σε πρώτο βαθμό τουλάχιστον. Γιατί αυτή η ιδέα δείχνει τουλάχιστον ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιτέλους κάτι άρχισε να κάνει σωστά. Δηλαδή, επιτέλους κατάλαβε ότι η ανταγωνιστικότητα είναι ο πυρήνος του θέματος για τη σταθερότητα της Ευρωζώνης και εκτός. Και συμφωνώ με τον Ιβάιλο ότι δεν είναι θέμα μόνο της Ευρωζώνης, πρέπει να αφορά όλη την Ένωση το θέμα αυτό. Όχι γιατί δεν μου αρέσει η Ευρώπη του ενός ή των δύο ταχυτήτων, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό. Θέλουμε σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα δύο συνδέονται τόσο στενά ώστε δίνεται να έχουμε σταθερότητα το ευρώ χωρίς να έχουμε σταθερότητα και των άλλων χωρών και αντίστροφα. Ακόμα και αν είναι μικρές. Θεωρώ λοιπόν ότι πρώτον χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες από τις κυβερνήσεις που προωθούν αυτή την πρόταση. Τι θέλουν να πετύχουν. Ακόμα δεν είναι σαφές. Και αν αυτό γίνει το Φεβρουάριο, έχουμε χρόνο μέχρι τις αρχές Μαρτίου να κάνουμε ένα ψήφισμα στο Ευρωκοινοβούλιο με τις απόψεις μας. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος ομιλητής ο κύριος Έγκλουντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι ένας από τους συγητές για το πακέτο της οικονομικής διακυβέρνησης έχουμε λέγει για το πακέτο αυτό και σχετίζεται με το θέμα που συζητάμε. Στην ομάδα των εισηγητών για το πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης ξεκίνησε το πακέτο αυτό το Σεπτέμβριο. Έγινε συζήτηση να συνδέσουμε με το πακέτο και τα άλλα θέματα έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε το πακέτο που έχουμε με την κανονική διαδικασία στο Κοινοβούλιο σαν μοχλό για να έχουμε ένα πούμε κάτι αν τυχόν το Συμβούλιο θελήσει ή δεν θελήσει να ε, μιλήσει μαζί μας. Πάντως έχουμε κακή εμπειρία όταν προσπαθούμε να συνδυάσουμε διάφορα, συνδέσουμε ορισμένα πράγματα. Πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι. Ορισμένες προτάσεις έχουν ήδη γίνει. Δουλεύουμε πάνω στο θέμα αυτό. για το πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης στην Οικονομική Επιτροπή. Έχουμε προθεσμίες. Αυτή τη βδομάδα λύγει η προθεσμία για τις τροπολογίες. Το δύσκολο στη συζήτηση είναι ότι συνεχώς συμβαίνουν νέα πράγματα. Το Συμβούλιο δουλεύει ουσιαστικά πάνω στο ίδιο πακέτο με εμά. Ταυτόχρονα όμως μερικοί πρωθυπουργοί όπως η κυρία Μέρκελ και άλλοι έχουν και δουλεύουν και ορισμένε νέες ιδέες που δεν έχουν ε, επίσημο χαρακτήρα γιατί δεν είναι το ίδιο οικονομικό, συγγνώμη, πακέτο για την οικονομική διακυβέρνηση που έχουμε εμεί στα χέρια μα. Και αυτό περιπλέκει τα πράγματα, γιατί οι δημοσιογράφοι, τα μέσα ενημέρωση, η συζήτηση στρέφεται γύρω από πράγματα που τυπικά δεν υπάρχουν. Ενώ έχουμε την άλλη μεριά με το πακέτο οικονομική διακυβέρνηση, την φυσιολογική διαδικασία εγώ λέω ας μείνουμε στη διαδικασία αυτή. Το έχουμε το πακέτο μεταξύ Συμβολίου και Κοινοβουλίου. Μερικοί εισηγητέ θα προσθέσουν επιπλέον στοιχεία που δεν υπήρχαν στην αρχική πρόταση της Κομισιόν, που μπορεί να διαφωνούμε με αυτά. Πάντως είναι στοιχεία που προσθέθηκαν εξωτερικά στο πακέτο που ήδη υπάρχει. Δεν θέλω φυσικά να μας ε, βάλουν στη γωνία κατά κάποιο τρόπο και να μην εξακολουθούμε να παίζουμε το ρόλο μα. Από μια άλλη μεριά δεν είναι εύκολα τα πράγματα ότι το Συμβούλιο κινείται προ 15 κατευθύνσει ταυτόχρονα. Το πακέτο οικονομική διακυβέρνηση, επαναλαμβάνω, αυτή τη βδομάδα έχει το πέραστο της προθεσμίας τροπολογιών. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ όλους σας. Μερικές παρατηρήσεις δικές μου. Όπως είπε ο εισηγητής και οι περισσότεροι συνάδελφοι που μίλησαν, πρέπει να δράσουμε γρήγορα, να πάρουμε μια γρήγορη απόφαση και η απόφασή μας πρέπει να είναι θετική. Άλλη επιλογή δεν έχουμε. Δεν μπορούμε συστηματικά να λέμε ότι ε, καθυστερούν να απαντήσουν οι κυβερνήσεις και τώρα να πούμε α, ε, ε, ε, αποφάσισαν υπερβολικά γρήγορα. Οι περισσότεροι συνάδελφοι ουσιαστικά συμφώνησαν με τους συζητητές μας. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με το έχουν τα πράγματα. Θα προτιμούσαμε ένα διαφορετικό μηχανισμό, πλήρως ευρωπαϊκό, κοινωτικό, Έχουμε όμως μια πολιτική κατάσταση τέτοια που είναι δύσκολο να κάνουμε κάτι άλλο. Εξάλλου στην πολιτική είναι υποχρεωμένο κανεί να λαμβάνει υπόψη την πραγματικότητα κάθε φορά. Όλοι οι συνάδελφοι έχουν καταλάβει ότι έχουμε τρεις κατηγορίες κειμένων. Έχουμε τη μήνυ συνθήκη, τη μικρή Τροπολόγηση της συνθήκης. Άρθρο 136. Αλλαγή του 136. Το Κοινοβούλιο εδώ μπορεί να δυσκολέψει το Συμβούλιο και μέχρι και αποτυχία μπορεί να οδηγήσει αν υιοθετήσει την απλή διαδικασία όπου είναι η, χρονοβόρα διαδικασία απαιτείται και μπορούμε να πούμε ουσιαστικά στην περίπτωση αυτή ότι τα μπλοκάρουν τα πράγματα. Μετά έχουμε το το πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης. Ο Σνάβος Σίγκλουντ είναι συνεισήγητη στην Οικονομική Επιτροπή έξι κείμενα. Και τρίτο, υπάρχουν διάφορες προτάσεις που έγιναν στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από ορισμένου πρωθυπουργού να συμπληρωθεί το σύμφωνο σταθερότητα με ένα σύμφωνο ανταγωνιστικότητα ή κάτι άλλο. και αυτό πρέπει να συζητηθεί, να το ξεκινήσει το θέμα να το μελετάει ο πρόεδρος Φαν Ρομπέι, η Κομισιόν, με στόχο το Μάρτιο. Με στόχο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να πετύχει μια συνολική συμφωνία το Μάρτιο. Έχοντας την ελπιζόμενη συμφωνία του Ευρωκοινοβουλίου και μια πολιτική συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με το πώς θα συμπληρωθεί το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Τρία διαφορετικά πράγματα. Εμείς εδώ είμαστε Επιτροπή Προπολογισμών. Το νομοθετικό πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης είναι πολύ ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι τη αρμοδιότητάς μα, με εξαίρεση ορισμένου από εσά που είστε μέλη στην Επιτροπή Οικονομική. Το ίδιο πράγμα για το Σύμφωνο ανταγωνιστικότητας. Και αυτό δεν είναι δικό μα χωράφι. Εμείς λοιπόν, εμάς μάλλον ως Επιτροπή Προβιζών μας αφορά το εξή. Αν είναι να συμβάλλει ο προπολογισμό της Ένωσης ή όπως συμβαίνει εδώ, αν αφού συμβάλλει ο προπολογισμό, θα πάψει να συμβάλλει. Αυτή την κατάσταση έχουμε μπροστά μας διότι ο μηχανισμός που εγκρίθηκε πέρσι στις 9 Μαΐου είχε ένα τμήμα διακυβερνητικό 440 δις και ένα κοινοτικό 60 δις με εγγύηση από τον κοινοτικό προπολογισμό. Ο νέος προπολογισμός, μη συγγνώμη μηχανισμός που θα τον αντικαταστήσει από το 2014 και μετά θα είναι 100% διακυβερνητικός καμία κοινωνική διάσταση. Διότι ορισμένες κυβερνήσεις και πιο συγκεκριμένα των χωρών που δεν είναι στην Ευρωζώνη και δεν σκοπεύουν να γίνουν σύντομα μέλη, δεν θέλουν να αναλάβουν κινδύνους έμεσα μέσω του κοινωνικού προπλοϊσμού να συμμετέχουν στη χρηματοδότηση του, του μηχανισμού. Το ερώτημα λοιπόν για μας, Επιτροπή Προπολογισμών, είναι μας ικανοποιεί το ότι ένα σύστημα προσωρινό μέχρι το 2013 που ξεκίνησε πέρυσι το Μάιο που είχε 60 δις κοινοτική διάσταση δάνεια με δεχόμενη εγγύηση από τον κοινότικό προπολισμό θα αντικατασταθεί από ένα σύστημα όπου ο κοινωνικός, ο κοινωνικός προπολισμός δεν θα υπάρχει πια. Και είναι λεπτό το θέμα για μας. Διασκεδαστικό θα έλεγα. Δηλαδή, εμείς είπαμε ναι για το μηχανισμό το Μάιο του 2010. Ταυτόχρονα όμως είπαμε ότι η εγγύηση που δίνει ο κοινωτικός προϋπολογισμός δεν χρηματοδοτείται ήταν ένα είδος πολιτική απόφαση με βάση την οποία οι κυβερνήσεις θεωρούσαν ότι η έμεση εγγύηση ήταν η διαφορά ανάμεσα στην οροφή των δημοσιονομικών προοπτικών και του ποσού του προεπλογισμού κατά κατηγορία, τι περιθώρια υπάρχουν σε σχέση με την οροφή, γιατί έτσι υπολογίστηκαν τα 60 δις. Αλλά αυτό ήταν τελείως θεωρία. Καμία νομική ισχύ δεν είχαν. Και το είπαμε εμείς αυτό. Και στα ψηφίσματά μας, Μπέγκε και λοιπά, είπαμε ότι στο ψήφισμα που θα ετοιμάσει η Επιτροπή ΣΟΥΡ θα πούμε ότι αν δοθεί διαρκής χαρακτήρα στο μηχανισμό αυτό θα πρέπει να βρεθεί ένα αντίβαρο, μια νομική οικονομική χρηματοδότηση για την εγγύηση αυτή εκ μέρους του προπολογισμού. Με το νέο μηχανισμό δεν τίθεται το θέμα αυτό πια. Αυτό είναι θετικό μεν για τον προπολογισμό μας που δεν απειλείται αλλά δεν είναι και πολύ καλό νέο για την κοινωτική πολιτική για την ευρωπαϊκή κοινωτική διάσταση, οικογενειακή θα την έλεγα, όσον αφορά τη χρηματοδότηση, τα οικονομικά μάλλον της Ένωσης. Από την άλλη μεριά έχουμε προθεσμίες. Οι εισηγητές μας είπαν ότι είναι πολύ βραχίας, βραχίας ορίζοντος. Πρέπει να γνωμοδοτήσουμε ως Επιτροπή και σας προτείνω γι' αυτό Πρώτον, να δούμε τι μπορεί να κάνει η Επιτροπή μας, η Επιτροπή Προϊσμών και τι χρονοδιάγραμμα. Θα αναφέρω το θέμα αυτό, θα το θέσω μάλλον στους συντονιστές, έτσι ώστε να δούμε από κοινού τι μορφή μπορεί να πάρει αυτή η κίνησή μας. Έχουμε χρόνο να κάνουμε γνωμοδότηση. Δική μας. Αν ναι, θα δούμε πότε. Αν όχι, Πώς μπορούμε να εκφράσουμε τη θέση μας. Βλέπω ότι υπάρχουν και διαφορετικές θέσεις. Υπάρχει όμως ταυτόχρονα και μια ευρεία ομοφωνία. Θα είναι επιστολή προς τον πρόεδρο, θα είναι μια τροπολογία που θα κατατεθεί από τις ομάδες μας. Ίσως είναι πιο εύκολο αυτό. Πρέπει να απαντήσουμε γρήγορα και ναι. Και όπως πολλοί από σας είπατε, θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία για το ψήφισμα τον Μάρτιο στην Λομέλια που θα είναι ένα συνολικό ψήφισμα για τη μεταρρύθμιση της ηθίκης και για τους έξι νόμους που σχετίζονται με την οικονομική διακυβέρνηση, έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να πει ποια θα είναι η θέση του. Εφ' Για τα, για τα κείμενα που θα έχουμε μπροστά μας σε λίγο καιρό, για τις προθεσμίες που θα έχουμε μπροστά μας και ενδεχομένως να ε, τροπολογήσουμε τη μεταρρύθμιση της ηθικής δηλαδή σε αντάλλαγμα το Κοινοβούλιο να πει ότι εφ' για όλες τις σημαντικές οικονομικές αποφάσεις είτε εξαρτώνται από την Επιτροπή Προπολογισμών, από την Επιτροπή Σούρη, από τη Συνταγματική, η ψήφο του Κοινοβουλίου θα εξαρτάται από και συμπληρώνουμε. Και ενδεχομένω να ζητήσουμε να πάρουν μέρο και τα Εθνικά Κοινοβούλια στην Οικονομική Διακυβέρνηση, Ευρωπαϊκό Εξάμεινο κλπ. Ξέροντα ο προπολογισμό μα, η Φραντζέσσα Μπαλτσάνη για τον προπολογισμό του 2012, που είναι το επόμενο σημείο, σκοπεύει να μας προτείνει το πώς προοδευτικά η συζήτηση για τον προπολογισμό για τον προπολογισμό της Ένωσης να μπει στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου Αυτό αφορά και τις δημοσιονομικές προοπτικές μετά το 2014. Συγητής Επιτροπής ΣΟΥΡ. Αυτά σας προτείνω αγαπητοί συνάδελφοι. Οι συγητές χρειάζονται ξανά το λόγο. Μάλλον όχι. Έλμαν. Ο Έλμερ δεν κοιμόταν, ε. Ζητάει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ρώτησαν κάτι μερικοί συνάδελφοι, γι' αυτό θέλω να πω σύντομα και την άποψή μου. Αλλά εσείς το περιορίσατε αντιστοίχως για την επιτροπή σας και η επιχειρηματολογία ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για δύο λόγους μπορεί να παίξει μόνο περιορισμένο ρόλο για το μηχανισμό στήριξης ε, έχει πρόβλημα όγκου έτσι, χρηματοδότησης. Γι' αυτό ο μηχανισμός στήριξης περνάει από τους εθνικούς ε, προϋπολογισμούς. Και υπάρχει και η ρήτρα για το no bail out, για τη μη διάσωση. Και για να αλλάξει αυτό δεν αρκεί μια απλουστευμένη διαδικασία για την τροποποίηση της συνθήκης. Και αυτό είναι θέμα των κρατών μελών και σχετισμού και πλειοψηφιών. Το δεύτερο όμως είναι αυτό που έθεσαν η κυρία Τρίπελ και ο κύριος Άλβαρο συμμετοχή των κοινοτικών θεσμικών οργάνων. Εγώ γι' αυτό μίλησα για τα θεσμικά όργανα συνειδητά και όχι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Διότι όντως σε πολλά θέματα δεν ε, απευθύνθηκε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη φάση. Ας πούμε για το πακέτο της ανταγωνιστικότητας και το αντίστοιχο σύμφωνο ανταγωνιστικότητας δεν είναι κατά κύριο ρόλο ε, αυτά θέματα ευρωπαϊκά. του μπορεί να ομοθετήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για συνταξιοδότηση και όρια ηλικίε κτλ. Και επίσης ε, τίθεται το θέμα ε, στην κοινοτική μέθοδο θα συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως τέτοια, ως όργανο ή μόνο η Γενική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, και γι' αυτό θα πρέπει να διαχωρίσουμε τα πακέτα. Το είπε και ο Πρόεδρος. Έχουμε τρεις διαφορετικές θεματικές ενότητες και πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Πρώτον, είναι αθέρωση συνθήκη. Και εκεί το όπλο μας δεν είναι το ε, θέμα της συναπόφασης, αλλά το χρονικό. Δεύτερον, έχουμε το Σύμφωνο Σταθερότητας και ανάπτυξη που και εκεί έχουμε συναπόφαση. Και τρίτον τώρα συζήτηση για το Σύμφωνο Ανταγωνιστικότητας, πλέον όπου δεν μας πέφτει λόγος καθόλου. Και ε, το θέμα είναι πού θα βάλουμε εμείς ακριβώς την προσπάθειά μας. Για να μην μας πετάξουν τελείως έξω, για να το πω, στα δύο από τα τρία πακέτα. Ακριβώς λοιπόν σε ποιο σημείο εμείς θα επέμβουμε ήδη από τώρα να χρησιμοποιήσουμε λίγο την τροποποίηση, την αναθεώρηση της συνθήκης για να παρέμβουμε, να αξιοποιήσουμε τις έστω και περιορισμένες δυνατότητές μας, όπως είπατε πρόεδρε, για να υπάρξει πολιτική δέσμευση του Συμβουλίου. Ή είναι καλύτερα να το κάνουμε στο στάδιο της νομοθετικής προετοιμασίας του συμβόλου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Και επειδή καταλήξαμε ότι δεν πάνε χρονικά και τα δύο παράλληλα, δεν θα πρέπει όμως να απεμπολίσουμε τα όπλα μας οι συνάδελφοι στην Οικονομική Επιτροπή δεν έχουν και καμιά τρομερή ιδέα για τις χρηματαγορές, ούτε για το θεσμικό οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό έχει χαλαρώσει λίγο στην αντίδρασή του και στο δυναμισμό του το κοινοβούλιο. Και δεν μπορούμε να σκεφτούμε και τα συνολικά ε, και τα υπερκείμενα. Και είναι ένα θέμα κύρους, επαναλαμβάνω, της Επιτροπής Προπολογισμών και αναγνώρισης και στάσεις. Και θα πρέπει να δούμε αν έχουμε το ανάστημα ε, και να το επιδείξουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν πρόκειται για σημαντικά θέματα. Εγώ δεν θέλω να είμαι κανένας Δον Κιχώτης εδώ, να κυνηγάω ανεμόμυλους, αλλά να ξέρουμε τι... Ε, αξιοπιστία έχουμε, γιατί αγωνιζόμαστε πολλές ε, περιπτώσεις να πετύχουμε συμβασμούς, μην χάσουμε κάθε κύρος. Για πρώτη φορά ευτυχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαστόματος του Προέδρου της είπε κάτι στο Κοινοβούλιο για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα ε, για τα χαρτιά, για την αναθεώρηση κτλ γιατί κυρίως για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται και κατά δεύτερο λόγο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα με ενδιαφέρε να ακούσω τι ε, θα γίνει με αυτά τα θέματα και πώς θα προχωρήσουμε. Τώρα δεν ξέρω εάν κατά πόσο τυπικά και επίσημα χρησιμοποιήσουμε την ενισχυμένη συνεργασία. Και μίλησαν και συνάδελφοι που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη χώρες τους. αν χρησιμοποιήσουμε de facto ή τύπη στην ενισχυμένη συνεργασία, σημαίνει αυτό ότι είναι σαφείς οι κανόνες βάσει των οποίων οι χώρες που δεν είναι μέλη του ευρώ έχουν ε, τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, να μην παραμένουν απ' έξω. Αυτό θα μπορούσε να είναι και έναυσμα, αν θέλετε, και κίνητρο για χώρες εκτός της Ευρωζώνης να μας βοηθήσουν λίγο. έτσι ώστε να μην αφήνουν τις χώρες Ευρωζώνης να τα θαλασσώνουν, να μας βοηθούν να βγάζουμε και πέρα. Θα μπορούσε και αυτό να είναι ένα σημείο συζήτησης και προβληματισμού τις επόμενες ημέρες. Παρακαλώ την άποψή σας. Και εσείς, Πρόεδρε, με τον τρόπο που σας χαρακτηρίζει, μπορείτε να βρείτε ένα τρόπο, δεν ξέρω τι διαδικασία, μια επιστολή ε, της Επιτροπής Προεπολογισμού που να διατρανώνει πραγματικά τη θέση της Επιτροπής σας. Αυτό θα βοηθούσε και τους δύο εισηγητές ε, της Συνταγματικής Επιτροπής. Θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμη μια τέτοια υποστήριξη της Επιτροπής σας για της επιστολής αυτής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σιγητά. Η Ίγκε θα να προσθέσει κάτι. Ναι, κυκλοφορεί μια φήμη ότι θέλουν και ξεχωριστό κοινοβούλιο τώρα, λέει, για τι χώρε τη Ευρωζώνη. Είναι μόνο φήμη ή ισχύει κάτι τέτοιο, έχει υπόσταση αυτό που ακούμε. Ε, κυκλοφορεί ναι, ένα έγγραφο από τη χώρα που γνωρίζω εγώ καλύτερα, όπως σας είπα προηγουμένως. Έχει τυπωθεί, αλλά είναι non-paper ε, αυτό το χαρτί, όπου ρητά γράφει ότι να υπάρχει μια συνέλευση των εθνικών κοινοβουλίων που να συνεδριάζει τακτικά για θέματα συμφώνου ανταγωνιστικότητας και για θέματα που είναι πέρα της εθνικής νομοθεσίας και το λέει αυτό το μη χαρτί μέσα. Μάλιστα. Πρόεδρε, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ για τις διευκρινίες και ευχαριστούμε τους δύο συνεισηγητές. Θα δούμε το θέμα αυτό στους συντονιστές ξανά σήμερα. Αγαπητοί συναδελφοί, ας περάσουμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Δυστυχώς, επειδή <clears throat> η ώρα περνάει, θα κόψουμε λίγο τα επόμενα σημεία. Αν και είναι μερικά σημαντικά, το 4 και το 5 για την προετοιμασία του προπολογισμού 12. Σας έχουν μοιραστεί τα έγγραφα. Θα σας τα παρουσιάσουν οι δύο εισηγητές. Δίνω αμέσως το λόγο στην Φρανσέσκα Μπαλσάνη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συναδελφοί, καταρχήν ευχαριστώ τη γραμματεία της Επιτροπής μας γιατί πραγματικά <clears throat> κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα και ακρίβεια. Είμαστε τυχεροί εμείς οι βουλευτές της Επιτροπής Προπλησμού που έχουμε τόσο πολύτιμη συνεργασία εκ μέρους της γραμματείας μας. <clears throat> Τώρα, ας συνεχίσουμε τη συζήτηση που είχαμε στις 26 του Ιανουαρίου όπου ε, εκφράστηκε η ανάγκη να ορίσουμε έναν πολιτικό προσανατολισμό για την έναρξη της διαδικασίας περπροϊσμού 2012 με πρόταση για ψήφισμα που θα σας την παρουσιάσω στη συνεδρίαση στις 3 Μαρτίου με αντικείμενο τη στρατηγική μας. για τη στρατηγική του... Συγγνώμη, για τον προπολογισμό 12. που συμπίτει με το πρώτο ευρωπαϊκό εξάμεινο, που γίνεται ένα κομμάτι δηλαδή της οικονομικής διακυβέρνησης και ένα σημαντικό εργαλείο για να πετύχουμε σε συνέργεια με τους εθνικούς προπολογισμούς το πρώτο βήμα για την, για την πολιτική στρατηγική 2020. Αυτό λοιπόν για την συνεδρίαση της Επιτροπής μας στις 3 Μαρτίου. Δυστυχώς το κείμενο θα το έχουμε μόνο στα αγγλικά και στα αγγλικά πρέπει να υποβληθούν και οι τροπολογίες λόγω έλλειψης χρόνου. Ελπίζω να συμφωνείτε. Έχω και ένα πρώτο χρονοδιάγραμμα για τις συναντήσεις με τις άλλες ειδικέ επιτροπές 28 Φεβρουαρίου μέχρι 22 Μαρτίου και που ελπίζουμε ότι θα μας βοηθήσουν στα πλαίσια της στρατηγικής 2020 να ορίσουμε τις προτεραιότητες που θέλουμε να δώσουμε εμείς στη δική μας ανάγνωση του προπολογισμού 2012. Έχετε πάρει το έγγραφο εργασίας. όπου εκφράζω καταρχήν, περιγράφω καταρχήν τη μέθοδο. Κάνω μια πρόταση πώς να επικαιροποιήσουμε την ιδέα αυτή του προπολογισμού με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο με βάση δύο σημεία. Μια προσπάθεια για διαφάνεια και καλύτερη κατανόηση του προπολογισμού για να τονίζονται ιδιαίτερα οι δαπάνες που είναι λειτουργικές και σχετίζονται άμεσα με τους στόχους του 2020, οι πέντε μεγάλοι στόχοι, και πέντε μεγάλες δράσεις, οι εφτά μεγάλες δράσεις και να συνδεθούν αυτές οι γραμμές του προπολογισμού του κοινοτικού με τους εθνικούς προπολογισμού. Θα έχουμε συνάντηση με τους εθνικούς βουλευτές στις 13 Απριλίου. Λειτουργικές δαπάνες, στρατηγική 2020, διαφάνεια και ενοποίηση κατά κάποιο τρόπο με τους εθνικούς προπολογισμούς. Βέβαια, ο πρώτος Λαμασούρ πέρυσι έκανε και αυτός ένα έγγραφο εργασίας για τη χρηματοδότηση της στρατηγικής 2020 μέσα σε συνθήκες κρίσης, προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η συνέργεια. Αυτά για τη μέθοδο. Μετά έχουμε τα νούμερα του προγραμματισμού. Κυρίως οι υποχρεώσεις. 147,12 δις ή 80 τόσο ανάλογα αν ληφθεί υπόψη το ε, Ταμείο ενίσχυσης. Αύξηση σχέση με τον προηγούμενο προπολογισμό 4,2%. Βέβαια, αυτή η αύξηση δεν είναι μεγάλη. Είναι εν μέρει φαινομενική, διότι εν μέρει οφείλεται στην ε, σχήμα χρηματοδότησης των ετησίων προγραμ... πολιετών προγραμμάτων που είναι διαφορετικά από χρόνο σε χρόνο Δεύτερον, η αυτόματη προσαρμογή 2%, μια ειδική αύξηση του 1β ως άμεση συνέπεια της αναθεώρησης όσον αφορά τις οροφές από την Κομισιόν και κυρίως μια μεγάλη αύξηση του κατηγορίας 2 που πρέπει να μειώνεται κάθε χρόνο. Μετά όμως είχαμε την, την, την επιστολή της Κομισιόν του Φθινοπόρου Οπότε ο λόγος της μείωσης των δαπανών σε σχέση με την αγορά γεωργικών προϊόντων είχα μεταβολή. Μετά μεγάλη αύξηση στο 2α λόγω των νέων οργανισμών και υπηρεσιών και όπως είπε και ο Πρόεδρος, κατηγορία 5 σε σχέση με την επιστολή Λεβαντόφσκη, Επιτρόπου Λεβαντόφσκη, που ζητάει να παραμείνει η αύξηση μέσα στα πλαίσια της οροφής 1%. Αυτά υποχρεώσεις πληρωμές δεν έχουμε νούμερα. Έχουμε μόνο την οροφή των δημοσιονομικών προοπτικών. 141,36 δις. Όπως έγινε και στο παρελθόν, μας ενδιαφέρουν τα περιθώρια. Μικρά περιθώρια, αλλά δεν είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που έλεγε ο προγραμματισμός πέρυσι. Έχουμε όμως μια πιθανή καινοτομία. Σε αντίθεση με το παρελθόν, φέτος μπορεί η πρόταση της Κομισιόν λόγω της κρίσης, της λιτότητας να είναι διαφορετική σε σχέση με, την, με τις προβλέψεις που είχαν γίνει. Να μείνει πιο χαμηλά δηλαδή ο αριθμός αυτός. Έχουμε ένα νέο σενάριο. Δηλαδή σημεία αναφορά στην πρόταση της Κομισιόν και τα περιθώρια να έχουν μία μεταβολή. Οπότε, το θέμα επίγει, μάλλον ορισμένα αιτήματα μπορεί να επίγουν. Πρώτον είναι οι μηχανισμοί ευελιξίας. Πώς θα χρησιμοποιηθούν. Οι συνήθεις μηχανισμοί αναθεώρηση των εγγραφών, το εργαλείο ε, ευελιξίας και η ευελιξία όσον αφορά το 5% που τώρα έχει νόημα προκειμένου να εφαρμοστούν προγράμματα που σχετίζονται στενά με τη στρατηγική 2020 αλλά και άλλα ερωτήματα που τα εγκαταλείψαμε καθοδόν όπως η ταυτοποίηση αρνητικών προτεραιοτήτων προγράμματα δηλαδή που θα μπορούσαν να χάσουν προτεραιότητα. Να οριστούν αρνητικές προτεραιότητες μπορεί να μας οδηγήσει σε απάντηση ότι δεν έχουμε αρνητικές προτεραιότητες, δεν θα γίνουν περικοπές. Έχει όμως νόημα παρόλα αυτά να θέσουμε το ερώτημα και υπεύθυνα να ακούσουμε την απάντηση αυτή. Στην προσπάθεια αυτή συνδυασμού ενός προπολογισμού λιτότητας με την ευθύνη που έχουμε ως ευρωπαϊκός προπολογισμό να βοηθάμε την οικονομική ανάπτυξη και στα κράτη-μέλη μας θέτει μπροστά σε ένα άλλο ερώτημα. Να ξεκινήσει δηλαδή μια συζήτηση για να βρεθούν νέα οικονομικά εργαλεία όπως η συμμετοχή της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Μια προσπάθεια για να συνδυαστεί η λιτότητα σε συνδυασμό με καινοτομίες, με όθεση της οικονομικής ανάπτυξης και προσπάθεια να καταπολεμήσουμε και εμείς την κρίση. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, παρακαλώ τον κύριο Φέρνανς που είναι εισηγητής για τα άλλα όργανα να μας πει και αυτό στη γνώμη του. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο προϋπολογισμός του 2012 καθώς και του 2013 θα είναι ε, προϋπολογισμοί κατά τους οποίους θα εδραιωθεί το νέο θεσμικό πλαίσιο και θα τεθούν και τα θεμέλια για την επόμενη προγραμματική περίοδο για τις δημοσιονομικές προοπτικές για ε, την καλή λειτουργία του Κοινοβουλίου και των λοιπόν θεσμικών όργανων. Αυτό που θα πρέπει να κυριαρχεί ε, στο μυαλό μας είναι και η αριστεία. Δεν θα πρέπει να συζητούμε μόνο για το κόστος της ε, μη Ευρώπης, της έλλειψης Ευρώπης, αλλά και το κόστος της έλλειψης αριστείας στην Ευρώπη. Θα πρέπει να ε, έχουμε στη διάθεσή μας τους πόρους, που είναι όμως απαραίτητοι για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει τα θεσμικά μας όργανα εδώ που έχουμε φτάσει να βασίζονται στην ε, χρηστή διαχείριση, ε, βεβαίως στην αποτελεσματικότητα αλλά και στην οικονομία και στην αριστεία. Αυτή είναι η στόχη μας και πολύ περιορισμένη η πόρη όπως γνωρίζετε. Και πρέπει να είμαστε σαφείς, απλοί, ε, με διαφάνεια, με αυστηρότητα στη διαχείρισή μας και όλα αυτά είναι στόχοι όχι μόνο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και για τα άλλα τμήματα και τα άλλα θεσμικά όργανα. Όπως θα δείτε και στην έκθεση, οι προσλήψεις θα γίνονται μόνο εφόσον έχουν εξαντληθεί δυνατότητες μετατάξεως προσωπικού, αξιοποίησης δηλαδή των υπαλλήλων που έχουμε ήδη. Επίσης, τα κτηριακά, ε, να δούμε ποια είναι τα πάγια έξοδα, ποια είναι τα ε, κείμενο με τα ε, έξοδα που μπορούμε να περιορίσουμε, να αποφύγουμε και πάντα βάσει αποτελέσματος να κρίνουμε. Ε, για να προχωρούμε πάντα με τρόπο σωστό και με περιορισμένους οικονομικούς πόρους. Θα πρέπει να υπάρχει και σωστός προγραμματισμός για το επόμενο πολιετές πλαίσιο, όπως σας είπα, να αρχίσει ήδη από τώρα. Γιατί έχουμε κάποιες πολιτικές ε, που δεν είναι πάντα πάγιες ή δαπάνες. Ε, παράδειγμα, η πολιτική της επικοινωνίας θα πρέπει να εκτείνεται σε περισσότερα έτη. Και για μια σειρά λοιπόν από πολιτικές, κάθε θητεία, στην αρχή της θητείας ε, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα άλλα θεσμικά όργανα καταρτίζουν ένα πρόγραμμα πολιετές για τον προϋπολογισμό τους. Πάντα με διαφάνεια. Και θα πρότεινα εγώ να ε, παρουσιάζεται στους ε, βουλευτές κάθε γραμμή του προϋπολογισμού ξεχωριστά και η εκτέλεση της, η πορεία της εκτέλεσης πολλές φορές στον χρόνο, όχι μόνο μία φορά το χρόνο, να παρακολουθούμε την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση, θα πρέπει πάντα να υπάρχει συντονισμός μεταξύ των διαφόρων θεσμικών ε, οργάνων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Και κάτι άλλο ένας άλλος τρόπος εξοικονόμησης χρημάτων για θέλετε είναι η καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που μας παρέχει η τεχνολογία. Ε, το, καλύτερη χρήση του ασύρματου διαδικτύου, ε, της ε, τηλεδιάσκεψης, της βίντεο διάσκεψης. Ήδη υπάρχει αυτός ο εξοπλισμός σε διάφορες αίθουσες και το ασύρματο διαδίκτυο και στα γραφεία των ε, ε, βουλευτών. Α, κάτι που ξέχασα είναι η πολιτική περιβάλλοντος, η είναι και στόχος 2020. Θα πρέπει να σεβαστούμε τις υποχρεώσεις και τις ε, ε, ενέργειες που μας αναλογούν. Ξέρετε ότι υπάρχει το σύστημα ΕΜΑΣ για οικονομία, εξοικονόμηση ενέργειας, χαρτιού, ε, αξιοποιώντας επαναλαμβάνω, τις ηλεκτρονικές δυνατότητες που έχουμε. Έτσι λοιπόν τα θεσμικά όργανα καλούνται να ε, ε, προτείνουν ε, που μπορούν να περικόψουν και να κάνουν οικονομίες στις δαπάνες τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ συνάδελφε. Επισημαίνω ότι ως προς το ζήτημα του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου, εκ της εκτιμήσεις δηλαδή για τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου, έχουμε ένα, μια δυσκολία το χρονοδιάγραμμα που θα πρέπει να διευθετήσουμε με το Προεδρείο. Θα πρότεινα να μην τη συστήσουμε τώρα στην Επιτροπή των Προπολογισμών, με τους συντονιστέ ε, μετά, αν θέλετε. Τώρα, αν θέλει, μπορεί να λάβει το λόγο η Συντόνια για να μας πει δύο λόγια. Μαζί με τη Φραντσέσκα είναι συν εισηγήτρια άλλου εγγράφου που σας έχει διανεμηθεί και που αφορά την υλοποίηση πιλωτικών προγραμμάτων και προπαρασκευαστικών δράσεων που βρίσκονται να εξελίξει Τόνια. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Όντως, σε συνεργασία με τη Φρανσέσικα, σήμερα παρουσιάζουμε ένα έγγραφο στην Επιτροπή που αποτελεί μία περιγραφή των πιλωτικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών δράσεων, τα όσα κάναμε στο Κοινοβούλιο και την Ολομέλεια το προηγούμενο φθινόπωρο. Τα πιλωτικά σχέδια δηλαδή και τις προπαρασκευαστικές δράσεις που έχει ε, εγκρίνει το Κοινοβούλιο, είτε πρόκειται για καινούργια σχέδια, είτε πρόκειται για παλαιότερα που παρατείνεται η ισχύ τους, η διάρκεια τους μάλλον. Και δεδομένου ότι δεν είχαμε την δυνατότητα πια το Δεκέμβριο Προσπαθώ με το έγγραφο αυτό για άλλη μια φορά να συνοψίσουμε αυτή την ε, δέσμη προτάσεων που τα είχαμε προτείνει στον προπολογισμό του 2011, το Δεκέμβριο που μας πέρασε. Στο παράρτημα υπαριθμών 1. Και προς ενημέρωση, στο παράρτημα 2 έχουμε μια απογραφή όλων των πιλωτικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών δράσεων που είχαν προβλεφθεί στον προπολογισμό του 2011 για να δείξουμε ακριβώς ότι δεν έχουμε αλλάξει τίποτα. Δεν έχουμε παρέμβει, απλώς καταγράφουμε τις ίδιες προτάσεις που είχαμε στο, στον αρχικό μας προπολογισμό. Θα δείτε επίσης νομική βάση για τις προπαρασκευαστικές δράσεις, για τα πιλωτικά σχέδια και πληροφορίες για όσους από εσά θέλουν να αναλάβουν μια τέτοια πρωτοβουλία προπαρασκευαστικού σχεδίου δράση. Επίσης έχουμε περιλάβει και ενημέρωση για τα όρια, τους περιορισμούς δηλαδή, που αντιμετωπίζουμε από την ε, συμφωνία και βέβαια από τα περιθώρια, που είναι πολύ σημαντικό πιστεύω να το σημειώσουμε. Να δείξουμε δηλαδή ποιο είναι το περιθώριο, ή μάλλον απουσία περιθωρίου ε, χειρισμών που έχουμε εμείς ως ε, συντάκτες. Και στο τέλος του εγγράφου θα δείτε ένα χρονοδιάγραμμα και εδώ θα ήθελα να υπογραμμίσω το εξής που είναι πολύ σημαντικό. Ως εισηγήτρια πέρσι διαπίστωσα ότι υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να αναλάβουν ε, τη διατύπωση ενός τέτοιου σχεδίου, πιλωτικού ή προπαρασκευαστικής δράσης και με χαρά βλέπουμε την υλοποίησή του. Όμως βλέπουμε ότι δυστυχώς ακόμη και οι ίδιοι οι προτείνοντες, οι συντάκτες των προτάσεων δεν δίνουν αρκετή προσοχή στα όσα πράγματι συμβαίνουν στην πρότασή τους. Υπήρξαν δηλαδή πιλωτικά σχέδια και προπαρασκευαστικές δράσεις που λησμονήθηκαν από τους ε, συντάκτες τους και τα οποία εγώ σκοπεύω βέβαια να παρακολουθήσω, να τα δω και φέτος με μέλημα κυρίως να δούμε αν υλοποιούνται οι στόχοι τους και επίσης εάν τυχόν αποτύχουν αυτές οι δράσεις ή τα σχέδια να ξέρουμε γιατί απέτυχαν. Να είναι πιο ξεκάθαρη δηλαδή η κατάσταση. Και επίσης στην υπόθεση αυτή αρρωγός μας στέκεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Συλλογή των Πληροφοριών. Στη σελίδα 5 του εγγράφου, παράγραφος 17, έχετε ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό, έχετε ενημέρωση για το πότε πρόκειται να κατατεθούν τα ε, οι προτάσεις για διορθώσεις. Και έχω να κάνω εγώ τώρα μια διευκρίνηση. Στην, ε, κατά την εβδομάδα υπαριθμών 16, περί της 20 Απριλίου αναφέρεται ότι θα συντάξει σχέδιο προϋπολογισμού η Επιτροπή και μαζί με αυτό θα καταθέσει πρόταση, ε, μάλλον έκθεση των πιλωτικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών δράσεων. Αυτό μάλλον θα καθυστερήσει. Θα έχουμε το σχέδιο μεν τον Απρίλιο, αλλά ε, συνοδευτικά έγγραφα και πρόταση για αξιολόγηση των πιλωτικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών δράσεων κατά πάσα πιθανότητα θα δούμε κάπου στις 25 Μαΐου από την Επιτροπή. Πάντως και με τη Φραντσέσκα Παρζάνη έχουμε υπόψη να ε, επικεντρωθούμε και σε μια από τις ομάδες ε, εποπτείας monitoring για αυτές τις ε, δράσεις και τα σχέδια και για το 2011 αλλά και μετέπειτα. Και γι' αυτό θα λάβω το θάρρος να συστήσω, εάν ενδιαφέρεστε, αν έχετε δηλαδή κάποια συγκεκριμένη ιδέα και θέλετε να κάνετε μια τέτοια πρόταση για πιλωτικό σχέδιο, ε, να το διαβάσετε να είστε ενήμεροι για το τι χρειάζεται, αλλά και γενικά αν θέλετε, αν σας ενδιαφέρει το θέμα αυτό και θέλετε να παρακολουθήσετε στο μέλλον τι γίνεται, να είστε ενήμεροι. Ευχαριστώ. Λέει η συγγετρία. Πολλοί συναδελφοί στον το λόγο. Παρακαλώ μια προσπάθεια όσο δυνατόν πιο σύντομα να εκθέσετε τις απόψεις. Ο κύριος Σούριαν είναι ο πρώτος. Ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ ιδιαίτερο την ε, συνάδελφο. Η Φραντσέσκα πέτυσε φόρο τιμή ε, στη γραμματεία μας, συνήθεια πολύ σωστή και καλή. Πρέπει και εγώ να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου, όχι μόνο γιατί είναι συνήθεια, αλλά για πολύ σοβαρό λόγο. Διαβάζοντα την πρόταση, πρέπει να πω ότι αρχικά αντιμετώπισα προβλήματα σε δύο επίπεδα. Καταρχά, δεν βλέπω, δεν έβλεπα μάλλον, δεν είδα χρονοδιάγραμμα σαφέ στη σχέση με τον προπολογισμό. Τώρα όμως, σε αυτή τη συνεδρίαση, έλαβα συμπληρωματικά έγγραφα που ε, αφορούν την συνεδρία των συντονιστών που θα λάβει χώρα αργότερα και εκεί είδαμε ικανοποίηση ότι προβλέπεται το χρονοδιάγραμμα και θα το συζητήσουμε. Ένα άλλο πρόβλημα για μένα το έγγραφο αυτό είναι ένα έγγραφο ε, σημαντικό και σε όγκο. Πλην όμως βλέπω ότι θα πρέπει η Επιτροπή μας και η Ολομέλεια στη συνέχεια να είναι εκείνες οι οποίες θα προσδιορίσουν τις προτεραιότητες για τον προπολογισμό. Από την παρέμβαση τώρα ακούω ότι η συγγήτρια είναι διατεθειμένη να ετοιμάσει ένα έγγραφο που θα έχει τις σχετικές προτάσεις όσο δεν με αφορά, ίσως ε, είναι αργά το να πούμε ότι θα ψηφιστεί το έγγραφο τον Απρίλιο, αλλά ίσως και να μην έχουμε άλλη ευκαιρία, δεν γνωρίζω. Ω προ την ουσία, η αύξηση 4,2% μου φαίνεται υπερβολικά φιλόδοξη, με δεδομένη την τρέχουσα κατάσταση. Βεβαίω το Συμβούλιο, όπω και την προηγούμενη χρονιά, διέπραξε το σφάλμα στις ε, πιστώσει ανάληψη υποχρεώσεων να είναι πολύ γενναιόδωρο και μετά στις ε, πιστώσεις πληρωμών να προσπαθήσει να είναι πιο ε, αυστηρό, να επιδείξει δημοσιονομική αυστηρότητα. Ίσως λοιπόν επαναληφθεί το ίδιο φαινόμενο και ίσως και για άλλη μια φορά, για άλλη μια χρονιά, να έχουμε σημαντική απόκληση μεταξύ των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών. Σε μια τέτοια περίπτωση, εγώ στηρίζω την συγκήτρια στην ε, πρόθεσή της, τη φιλοδοξία της να επιδείξει θάρρος και παρησία και να υψώσει το ανάστημα ως προς τα ε, θέματα των αρνητικών προτεραιοτήτων. Γιατί συμφέρον του Κοινοβουλίου και φαντάζομαι και του Ευρωπαίου πολίτη είναι ο προϋπολογισμός, ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός να εξυπηρετεί ακριβώς τις ανάγκες του πολίτη. Εάν ε, υποχωρήσουμε σε κάθε σημείο, ο προπολογισμό δεν θα αποστέλει κανένα μήνυμα στον πολίτη. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα σημαντικά, στι αυξήσει που θεωρούμε πιο σημαντικέ και τι δαπάνε μα να τι εστιάσουμε ακριβώ στου τομεί αυτού. Και εδώ χρειαζόμαστε συνεργασία και βέβαια σύμπραξη στη ψηφοφορία για να έχουμε τι απαραίτητε πλειοψηφίε. Επίση, πολύ σημαντικό θα ήταν να συνεχιστούν οι προσπάθειες με βάση τις ιδέες για τους νέους ίδιους πόρους. Και ίσως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, να αποτελέσει τη λύση αυτή που άλλωστε ε, υποστηρίζει εδώ και καιρό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να συμπεριληφθεί δηλαδή και εκείνη. Ξέρουμε βέβαια ότι το Συμβούλιο αντιδρά με προϋπόθεση ε, λέγοντα ότι ναι, μπορεί να γίνει, αλλά η προπόθεση είναι να μην αυξηθεί το συνολικό ποσό, η η συνολική επικοδότηση του προπολογισμού. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει από αλλού να, βρουν, βρεθούν τα κονδύλια για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πράγμα αδύνατον. Εάν αυτό εννοούσε η εισηγήτρια ω ε, συνεργασία, ε, εάν θεωρείτε ότι υπάρχουν άλλε εναλλακτικέ, μακάρι, τι να πω. Αλλά για τον προπολογισμό του 2012 δεν βλέπω άλλε λύσει πιθανέ. Και μια τελευταία παρατήρηση, Πρόεδρε φρονώ ότι πρέπει πάντοτε να στηρίζουμε τα, μακρόπνοα, τα μακρόπνοα σχέδια που έστω και αν δεν είναι επίκαιρα, αν δεν είναι ενημερωμένα στις τρέψεις κινήσεις οι συνθήκες, μπορούν να αποτελέσουν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούμε, μέσα στο οποίο θα βρούμε τους διάβλους για την πρόοδό μας, αλλά και για τη συνεργασία μας. Και γι' αυτό θα ήθελα να δω νέες προτάσεις για νέες προτεραιότητες, Πέρυσι είχαμε θέσει ως επίκεντρο της προσοχής μας την νεολαία. Φέτος περιμένουμε πάλι ένα μεγάλο σχέδιο, ένα όραμα το οποίο να μπορούμε όλοι να στηρίξουμε και με αυτό να αποστείλουμε ένα σεφές μήνυμα στον Ευρωπαίο πολίτη. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Εγκλούτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω ε, την εισηγήτρια μας και την βασινή εισηγήτρια και ε, σε ό,τι αφορά το κοινό ψήφισμα, ε, όπως είχαμε συζητήσει και σε προηγούμενη συνεδρίαση, συμφωνώ με την προσέγγιση. Επιτρέψτε μου επίσης να πω ότι δεν συλλεύω καθόλου την κυρία Παρζάνη που είναι η συγγήτρια για το 2012. Γνωρίζουμε πόσο δεν είναι η οικονομική κατάσταση και yeah. Ε, αν θεωρήσουμε ότι ήταν δύσκολη στη διαπραγματεύση για τον προπολογισμό του 2011, πόσο μάλλον του 12. Ε, είναι και τα περιθώρια πάρα πολύ στενά. Όπως είπαμε, η κατάσταση είναι δύσκολη. Εγώ μελέτησα πάρα πολύ προσεκτικά το έγγραφο θέσεων της συγγητρίας και πάλι βρίσκω ενδιαφέρον αυτό που λέει για το πώς θα ενταχθεί στο προϋπολογισμό η ιδέα της οικονομικής διακυβέρνησης, economic ε, governance. Ε, και είναι ενδιαφέροντα αυτά που λένε και οι εθνικές κυβερνήσεις και το Συμβούλιο, αλλά σε θεωρητικό επίπεδο και παραμένουμε πολύ στο θεωρητικό επίπεδο. Τι θα γίνει τώρα στο διατάφτα. Πώς θα τα εφαρμόσουμε όλα αυτά στην πράξη. Εγώ δεν το έχω ξεκαθαρίσει ακόμα. Ακόμα και αν διάβασα το έγγραφο προσεκτικά, το έχω πει και σε προηγούμενη συνεδρίαση. και εισηγητή στην Οικονομική Επιτροπή για αυτό το θέμα της οικονομικής διακυβέρνησης, όπου έχει μάλλον περιορισμένο, περιθωριακό ρόλο ο κοινοτικός προϋπολογισμός σε αυτή τη συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή. Τώρα σε τι ανάγεται αυτή η συζήτηση, ρωτάτε κι εσείς, αν θα πρέπει να έχουμε αρνητικές προτεραιότητες. Αυτά τα λέει και η Επιτροπή Σούρε. Είναι πιο δύσκολο να έχει κανείς αρνητικές προτεραιότητες στο πλαίσιο των πολιετών δημοσιονομικών προοπτικών. Είναι πολύ δύσκολο από τώρα ε, να βρεθούν πόροι στον ε, προπολογισμό, αλλά ταυτόχρονα είναι επιτακτική ανάγκη να απαντηθούν ε, ορισμένα ζητήματα και το Συμβούλιο τώρα καλεί για ολόκληρο σύμφωνο ανταγωνιστικότητας. Μα αν δεν μπορούμε να έχουμε προτεραιότητα, α πούμε, την εφαρμογή της στρατηγική του 2020 με ανακατάταξη και αναθεώρηση των προτεραιοτήτων στον προπολογισμό για να βρούμε και φρέσκο χρήμα. Αν δεν κάνουμε τίποτα το 12 και το 13, έχει πάει χαμένο ουσιαστικά ε, ο χρόνος, το τρίτο του χρόνου που είχαμε στη διάθεσή μας. Όταν αρχίσαμε αυτή τη συζήτηση για το 2020 ήταν 10 χρόνια πριν. Και αν λοιπόν ε, πάνε στο βρόντο τώρα το 12 και το 13 θα έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος, το, 30% του χρόνου. Δεν είναι εύκολο από τώρα να δούμε κάποια ζητήματα για τις ε, δημοσιονομικές προοπτικές, αλλά ίσως πρέπει να συζητήσουμε κάποιες αρνητικές προτεραιότητες ε, για να τονιστούν και οι θετικές μας, οι πραγματικές. Αν θεωρείτε ότι μπορεί να βρεθεί ισορροπία ανάμεσα στην εξηγίαση των δημοσίων οικονομικών και εξέβρεση πόρων για επενδύσεις παραγωγικές για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγικότητας, ε, ακριβώς αυτό είναι η χρυσή τομή. Ε, δεν ξέρω αν είναι δυνατόν, πρέπει να είναι δυνατόν, αλλά ακριβώς να εντοπιστούν οι αρνητικές προτεραιότητες. Εύκολο δεν θα είναι να φτάσουμε σε μεγάλο περιθώριο για τον προπολογισμό πέσει, καταφέραμε να φτάσουμε το 2,97% του χρόνου, δεν ξέρω. Εκτός αν περισσέψουν κάποιοι πόροι στα διαρθωτικά ταμεία ή στην έρευνα για να έχουμε ένα περιθώριο χειρισμών, αν υπάρξει ευελιξία. Αυτό όμως εναπόκειται και στο Συμβούλιο για τη χρηματοδότηση άλλων στόχων και άλλων προτεραιοτήτων. Μένει να αποδειχτεί αυτό. Εγώ με μεγάλη μου χαρά προσβλέπω στη συνεργασία και στο τελικό ψήφισμα θα παρακολουθήσω την όλη διαδικασία αυτή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ αγαπητές συνάδελφοι. Ο Γεραν Φέρμ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να κάνω μερικά σχόλια και για τις δύο εκθέσεις των δύο εισηγητριών. Πρώτο για την έκθεση Βαλσάνη. Για το γενικό προϋπολογισμό. έκανε μία μεθοδολογική πρόταση για το ψήφισμα. Συμφωνώ. Να είναι πάρα πολύ συνεκτικό και εστιασμένο. Και επίσης πολύ καλή ιδέα για το έγγραφο που έχει κάνει αυτό εδώ το έγγραφο για τη στρατηγική που να βασίζεται στο δημοσιονομικό προγραμματισμό. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Βλέπουμε κάποια σημεία που θα είναι προβληματικά και χρειάζεται ανάλυση καλή. Είναι προφανές θα είμαι πολύ σύντομος. Είναι προφανές ότι η στάση και η συμπεριφορά του Συμβουλίου θα ε, μας προκαλέσει κάποια προβλήματα. Το είπε και ο Έγκλουντ. Πώς θα βρούμε την ε, ισορροπία ανάμεσα στη λιτότητα και την οικονομική ανάπτυξη και τι ρόλο μπορεί να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διερευνήσουμε λίγο περισσότερο ορισμένα θέματα. Θα πρέπει να δώσουμε στο Συμβούλιο να καταλάβει ότι ο προϋπολογισμός βασίζεται σε κάποια προγράμματα ε, πολυετή που είναι και νομικά δεσμευτικά. Σε αυτό βασίζεται ο προϋπολογισμός ο ίδιος, είναι η ίδια βάση. Δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε, να τα παρακάμψουμε, να τα παραγωνίσουμε, να το χωνέψει αυτό το Συμβούλιο. Επίσης η ανάληψη υποχρεώσεων είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να πληρώνεται. Δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει ε, πέρυσι αρχίσαμε να μειώνουμε το χάσμα, να κλείνουμε την ψαλίδα ανάληψη ε, υποχρεώσεων και πληρωμών. Θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η τάση, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να δούμε πώς θα γίνει αυτό, πώς θα συμφωνήσει το Συμβούλιο. Χρειάζονται πάρα πολύ καλά επιχειρήματα. Αλλιώς θα αφήσουμε μεγάλες περιφέρειες και σημαντικά προγράμματα στα κρύα του λουτρού. Τα χρήματα αυτά έχουν υπολογίσει. Ε, είναι και ένα θέμα αναδιανομής του πλούτου, ε, αλληλεγγύης. Παίρνουμε από τους πλουσίους και δίνουμε στους φτωχούς. Δεν κερδίζουν όλα τα κράτη-μέλη από τις περικοπές στον προϋπολογισμό. Ε, ορισμένα κράτη και συγκεκριμένα περιφέρειες χάνουν από τις περικοπές του κοινοτικού προϋπολογισμού. Δεν ξέρω αν τα βλέπει αυτά το Συμβούλιο. Και κάτι άλλο. Αν δεν μπορέσουμε Μάλλον, για να το εξηγήσουμε αυτό στο Συμβούλιο, χρειαζόμαστε υποστήριξη των ε, επιμέρους ειδικών επιτροπών για ε, τα νομοθετικά προγράμματα, τα πολιετή, για να βρούμε, να αντλήσουμε από εκεί τα ε, απαραίτητα επιχειρήματα και να μπορέσουμε να πείσουμε με στένος το Συμβούλιο. Αυτά για την έκθεση κυρίας Μπαρζάνη που είναι πολύ καλά και πολύ χρήσιμα. Έρχομαι τώρα στην άλλη έκθεση τώρα του κυρίου Φερνάντες, πολύ καλή, ε, ίσως λίγο πιο παραδοσιακή. Μου λείπουν μερικά στοιχεία όμως. Πρώτον, έχουμε ζητήσει από το ε, Προεδρείο και άλλα όργανα καμιά φορά για περισσότερη ενημέρωση ε, εκθέσεις για προπολογισμό από μηδενική βάση, τις διάφορες ε, μεταβλητές, τις διάφορες δαπάνες, πάγιες ή μη, ε, για τον οίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, για τα κτίρια, όλα αυτά τι κοστίζουν. Τώρα φτάνουμε στο στάδιο των συμπερασμάτων και δεν βλέπω πάρα πολλά συμπεράσματα στην έκθεση αυτή. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε και σε αυτά τα πολύ επίμαχα θέματα. Τι θα το κάνουμε το κέντρο των επισκεπτών, τον οίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, το καθεστώ των βοηθών μας και το πιο δύσκολο από όλα, ίσως, είδαμε την επιστολή του κυρίου Λεβαντόφσκι που μας ζητεί να περιορίσουμε την αύξηση στο 1% ονομαστικά, έτσι, που σημαίνει ουσιαστικά με πραγματικούς όρους περικοπή. Όταν αφορά αυτό το προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου, εμεί πώς θα απαντήσουμε και τα άλλα θεσμικά όργανα πώς απαντούν. Για μας βεβαίως είναι ε, θέμα του προπολογισμού του Κοινοβουλίου και θα πρέπει να μας απασχολεί στη μελλοντική συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χάρτονγκ. Eh, eh, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να αντιδράσω ε, για την έκθεση κυρίας Βαρζάνη και της Ιδονίας. Νομίζω εδώ βρήθη ε, διαφόρων πιλωτικών ε, προγραμμάτων. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φέρει την έκθεση εφαρμογής για να ελέγχουμε γιατί και αυτή είναι η δουλειά μας ε, ως βουλευτές, ότι τα προγράμματα είναι σωστά, αποτελεσματικά και πιάνουν τόπο. Για την άλλη έκθεση, για το 2012, ποια είναι η πραγματική πολιτική ε, ε, για τον προπολογισμό. Λυπάμαι που δεν βλέπω περικοπές, εξοικονόμηση και δεν έχει γίνει δυστυχώς η μάχη που έγινε πέρσι και λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό, κυρίως για τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφοι. Η Έλγα, Τρούπερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους δύο εισηγητές. Στα αγγλικά, κυρία Τρούπελ, θα αρχίσω από τη Φραντσέσκα. Ε, γνωρίζεις ότι είμαι μέλος των Πρασίνων και ως μέλος των Πρασίνων είμαι πάρα πολύ ε, ε, μεγάλη υποστηρίκτρια του εξυγχρονισμού της Ένωσης μέχρι το 2020 και αν εφαρμόζεται σωστά η στρατηγική αυτή μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη. Έρχομαι τώρα στη συγκρούση των στόχων στις εμβληματικές ε, ε, πρωτοβουλίες ε, αναφέρονται οι πόροι για μια καλύτερη Ευρώπη, αλλά στη γεωργία και στις διαρθρωτικές πολιτικές χρειάζονται για να υπάρξουν πραγματικές προτεραιότητες αλλαγές και στον προπολογισμό της συνοχής για περισσότερη αηφορία και ε, εξοικονόμηση των πόρων, αποτελεσματική χρήση. Και το πρόβλημα που έχουμε εκεί δεν είναι μόνο ε, πρόβλημα του Συμβουλίου, αλλά και τον συσχετισμό και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι νέε πλειοψηφίε δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα. Αν δείτε τι ισχύει και στι ψηφοφορίε τη Επιτροπή ΣΟΥΡΕ. Μα αν θέλουμε νέε προτεραιότητε, κάπου πρέπει να περικόψουμε παλιέ προτεραιότητε. Γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν θα αυξηθεί σημαντικά ο υπολογισμό. Δεν είναι ρεαλιστικό αυτό. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι να τα ρίχνουμε όλα στο Συμβούλιο. Έχουμε και εμεί εσωτερικά προβλήματα. Και αν δεν είμαστε έτοιμοι να ε, βρούμε νέες προτεραιότητες, θα έχουμε πάνω κάτω τον παλιό προπολογισμό με τα παλιά προβλήματα. Αυτό είναι ο κίνδυνος που διαβλέπω εγώ. Έρχομαι τώρα στην έκθεση του κυρίου Φερνάντες. Γενικά, ο στόχος ε, της εξυγίανσης είναι πολύ ωραίος και καλός. Αλλά εγώ δεν βλέπω τις λεπτομέρειες εδώ ε, στο γενικό τίτλο που αναφέρεται. Διότι το μόνο που ακούμε είναι ότι θέλετε να ε, επενδύσετε περισσότερο στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, στο ασύρματο διαδίκτυο και ε, στη υπόθεση του περιβάλλοντος. Και μετά λέτε για οικονομίες. Δηλαδή πρώτα να επενδύσουμε σε αυτές τις τεχνολογίες και μετά να κάνουμε οικονομίες. Για τον οίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας ακούσαμε. Δεν ξέρω, δεν βλέπω πουθενά πώς θα μπορέσετε να το χρηματοδοτήσετε σύμφωνα με την εξηγίαση και αν ε, είστε σοβαροί σε αυτή την πρόταση. Και εσείς και το ΕΛΚ τώρα δεν θα πρέπει να πάτε σε μια δεύτερη φάση ε, ε, για το καθεστώς των βοηθών. Από πέρσι είχαμε συγκρουστεί για αυτή την υπόθεση. Μάλλον θα πρέπει να τα να θεωρήσετε αυτά, γιατί δεν καταλαβαίνω αυτά που λέτε για την εξηγήση του προπολογισμού ε, γενικά και αόριστα, ε, αν δεν μας προτείνετε συγκεκριμένα πού θα βρείτε τα χρήματα αυτά. Ευχαριστώ. Πολύ εύστοχη παρατήρηση και η Αΐντερ Γόρδια Σάμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα, γιατί μίλησαν πολύ. Ιδιαίτερα ε, για το έγγραφο της κυρίας Βαρσάνη. Θα ήθελα να τη συγχαρώ. Συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό και στις απόψεις μας και στον τρόπο προσέγγισης του επόμενου προπολογισμού. Έτσι κι αλλιώς θα χρειαστεί βοήθεια η συγκήτρια, το γνωρίζουμε όλοι. Κάνει ε, κάποιες προτάσεις και κάποιες ερωτήσεις θέτει στο κείμενό της και νομίζω ότι ήδη μπορούμε να αρχίσουμε να τις απαντάμε. Ο κύριος Φέρμα απάντησε ήδη για τις πληρωμές. Τι επίπεδο πληρωμών θα πρέπει να ε, επιζητούμε ή να, να υπερασπιζόμαστε. Πρώτα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει περισσότερα στοιχεία, να καταθέσει αντίστοιχη πρόταση σε ένα κείμενο, να βλέπουμε ποιες είναι οι πληρωμές, ε, ανταποκρινόμενες στις ε, υποχρεώσεις που ήδη έχουμε αναλάβει. Το λέει και η συγγήτρια ότι αυτά είναι δεδομένα. Πάντως, καταρχήν αυτό δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Αυτό που εμείς θα πρέπει να υπερασπιζόμαστε θα πρέπει να είναι η ανάληψη υποχρεώσεων οι πληρωμές απορρέουν από ε, τους κανονισμούς για την εκτέλεση των προγραμμάτων. Το Συμβούλιο μπορεί να κάνει μια σωστή ή λανθασμένη ανάγνωση αυτών, ε, επειδή θέλει ή έχει φιλοδοξίες περικοπών. Δεν χρειάζεται εμεί να έχουμε την ίδια στρατηγική. Έχουμε μια στάση στη διαπραγμάτευση Δεν ξέρω αν θέλετε τώρα αντί να υπερασπιζόμαστε την ανάληψη υποχρεώσεων, να έρθουμε να υπερασπιστούμε τις πληρωμές, να έχουμε ένα ελάχιστο όριο πληρωμών, ένα αυτό θα πρέπει να το δούμε. Ε, ρωτάει τώρα η κυρία Μαρσάνη για τις ανετικές προτεραιότητες. Αυτό είναι πολύ σημαντική άσκηση. Όχι λόγω τη κρίση, αυτό κανονικά θα έπρεπε να έχει γίνει, γιατί και εγώ είμαι καινούριο βουλευτή εδώ, θα πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο. Υπάρχουν κάποια προγράμματα που τρέχουν, ε, που αποδίδουν και χρειάζεται να επενδύσουμε σε αυτά. Εάν δεν πηγαίνουν καλά και δεν μπορούν να βελτιωθούν, να τα καταργήσουμε. Όχι λόγω κρίση. αυτό πρέπει να είναι πάγιο. Άλλο είναι η κρίση. Αν είναι κρίση και περιορισμένο ο προπολογισμό με περικοπέ κτλ που δεν είναι και δεδομένο, θα πρέπει να αγωνιστούμε γι' αυτό, που θα πρέπει να γίνουν περικοπέ. Ε, από εκεί και πέρα αρχίζουμε και συζητάμε για προτεραιότητε, μεγαλύτερε ή μικρότερε. Για τι αρνητικέ, ό,τι δεν πάει καλά θα πρέπει να το εξετάζουμε, είτε έχουμε κρίση, είτε επέκταση οικονομία. Δεν κατάλαβα. Τα χρήματα που αντλούμε από τον κοινοτικό προπολογισμό θα πρέπει να πιάνουν τόπο, να την χάνουν χρηστή διαχείριση. Δεν το λέω για την κυρία Βασάνη καθόλου σε καμία περίπτωση, αλλά φαίνεται ορισμένοι τα σκέφτονται αυτά μόνο σε περίοδου ε, κρίση. Επίση κάνει λόγο για τη χρήση του μέσου ευελιξία, κυρίω για την κατηγορία 1α και την κατηγορία 4, που ξέρουμε ότι εκεί κυρίω είναι τα προβλήματα. Και αφού είναι τόσο περιορισμένα τα περιθώρια και το περιθώριο του προπολογισμού και το περιθώριο ρηγμό, θα πρέπει να καταφύγουμε. Τι να κάνουμε ε, στο μέσο ευελιξίας. Για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ξέρετε πόσες φορές τα έχω ακούσει. Πανάκια, το τελευταίο χρόνο όλο γι' αυτό ακούω και στη Σούρε και εδώ. Βεβαίω είναι σαφέ ότι θα πρέπει να συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και να βοηθήσει να φτάσουμε στου στόχου μα. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον προπολογισμό και το μερίδιο που μα αναλογεί. Αν θέλετε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την Τράπεζα Επενδύσεων ε, ως συμπληρωματική τη δική μα δράση, όχι ω πρόφαση για να κάνουμε περικοπέ στο δικό μα προπολογισμό. Merci, Πολλοί ακόμα έχουν ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ να είστε σύντομοι. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήσει. Η μία αφορά τον προπολογισμό του Κοινοβουλίου και νομίζω ότι πια είναι η ώρα να καταστήσουμε σαφέ στην κοινή γνώμη ότι κάνουμε και εμεί προσπάθειε για λιτότητα. Και αν δούμε τα στοιχεία του 2010, 75 ήταν οι θέσει για το Κοινοβούλιο με βάση την ε, Λισαβόνα και 430 ήταν αυτές που εξασφάλισε η Γραμματεία. Εδώ λοιπόν είναι πολλά πράγματα στα οποία θα μπορούσαμε να πείσουμε, να δείξουμε στον κόσμο ότι έχουμε καταφέρει πολλά πράγματα και ε, ότι αγωνιζόμαστε ακόμη και απέναντι στο ε, Προεδρείο του Κοινοβουλίου. Είναι πολλά τα σημεία στα οποία μπορούμε πράγματι να εξοικονομήσουμε χρήματα και μακροπρόθεσμα μάλιστα. οι δύο πρόσθετες εβδομάδες αργιών για τους, ε, για τους εργαζομένους ήδη είναι ένα πολύ καλό ε, δείγμα που θα μπορούσαμε να ε, προβάλλουμε. Για τα πιλωτικά σχέδια και τις επανασκευαστικές δράσεις θα μπορούσαμε να πούμε ναι, ότι μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα και να εξασφαλίσουμε τα 15 εκατομμύρια. Αλλά το θέμα είναι αλλάζουμε τα περιθώρια και μπορούμε να στήσουμε από το Συμβούλιο και άλλα χρήματα. Θα ήθελα οι συνάδελφοι να μου πούνε τι γνώμη έχουν για την υπόθεση αυτή, πώ θα μπορούσαμε να σταθούμε δηλαδή απέναντι στην Επιτροπή και το Συμβούλιο. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Πολύ σημαντικό. Κύριο Άλβαρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα σταθώ στην έκθεση του κυρίου Φερνάντε για να πω ότι πρέπει οπωσδήποτε να ε, υποστηρίξουμε τις, και να επιδιώξουμε τις αρχές της αποτελεσματικότητας, διαφάνειας, του ελέγχου, της βιωσιμότητας, όπως η παραδείγμα της προτάσεις περί περιορισμού της ε, χρήσης χάρτου, της κατανάλωσης χάρτου. Νομίζω ότι είναι σοβαρό θέμα, μπορούμε να περιορίσουμε Φερρυπίν τον όγκο του χαρτιού μόνο και μόνο καταργώντα τη μία από τι δύο αποστολέ ημερήσια διάταξη τη συνεδρία. Δεν χρειάζεται να φεύγει και με το εσωτερικό ταχυδρομείο ημερήσια διάταξη και να την ε, παίρνουμε στην ε, είσοδο τη αίθουσα. Επίση, θα ήθελα να επισημάνω, όπω είπε και η κυρία Τρίπελ, ότι πολλά είναι θετικά στοιχεία στην προσέγγιση αλλά στην υλοποίηση. Τελικά λείπουν κάποια ε, στοιχεία για να εξασφαλίσουμε περισσότερη αποτελεσματικότητα. Στο σημείο M, επί παραδείγματι, οι προτεραιότητες σε σχέση με τα κτίρια που πρόκειται να ενοικιαστούν. Και νομίζω ότι εδώ μπορούμε να συζητήσουμε υπενθυμίζοντας ότι και η Επιτροπή αναζητά ε, ένα τέτοιο κτίριο και ότι προσπαθούμε να αποφύγουμε μια υπερβολικά δαπανηρή ε, διαδικασία για ε, μίσθωση κτηρίου ε, που δεν προβλέπει προαίρεση εξώνησης. Επίσης, σε θέματα φερειπίν της Επιτροπής Περιβάλλοντος και συνοπολιτισμού και επικοινωνίας, επικοινωνιακής πολιτικής η στάση την οποία θα τηρήσουμε και η αποτελεσματικότητα στις επιλογές μας νομίζω έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και πιστεύω ότι ήταν ε, δυσάρεστη η έκπληξη, η έκπληξη που είδαμε ε, στην Επιτροπή Πολιτισμού όταν ε, διαπιστώσαμε ότι ο προϋπολογισμός μας για το 2012 μάλλον θα έχει διαφορετική πρηγοδότηση από ό,τι περιμέναμε. Επίσης θα πρέπει να δούμε το προσωπικό. Το 2012 πρόκειται να αυξηθεί, πρόκειται να ενισχυθεί. Η γραμματεία του Κοινοβουλίου θα προσλάβει, η Γενική Γραμματεία θα προσλάβει περισσότερο προσωπικό και με ποιο σκοπό, τι χρήση θα έχει αυτό το προσωπικό. Άκουσα διάφορες φήμες, που δεν ξέρω αν είναι βέβαια βάσιμες, ότι υπάρχουν κάποια, κάποιες τάσεις ή συμφέροντα σε επίπεδο γραμματείας του Κοινοβουλίου, να ενισχυθεί πολύ το, το γραφείο του Προέδρου, το επιτελείο του Προέδρου, ώστε να μπορεί να αναλαμβάνει και έργο το οποίο δεν σχετίζεται άμεσα με την καθοδήγηση των εργασιών του Κοινοβουλίου και με τον κανονισμό. Επίσης, Σημαντικό, όπως είπε και ο κύριος Φέρμ, είναι να έχουμε την αξιολόγηση, τον υπολογισμό του κόστους ε, και του ωφέλους. Να δούμε δηλαδή ουσιαστικά τι κερδίζουμε στο σημείο 12. Με τις ε, <coughs> θέσεις εργασίας ε, περιορισμένου χρόνου ή με τις ε, βίντεο διασκέψεις. Τι μας προσφέρουν όλα αυτά. Μπορούμε, Φερρυπή, να κάνουμε εξοικονόμηση κονδυλίων σε σχέση με τις αποστολές των αντιπροσωπιών μας. Μετά, κάτι άλλο που δεν απαριθμείται εδώ, αλλά είναι πάρα πολύ επίκαιρο ενδεχομένω ως θέμα, είναι το εξή. Θα πρέπει να κοιτάξουμε αν δαπανούμε σωστά ε, τα κονδύλια για την ασφάλεια. Όποιο ήταν εδώ την Παρασκευή θα κατάλαβε ότι για τρίτη φορά φέτος, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ε, πώς να το πω, καταργήθηκε, ακυρώθηκε το σύστημα ασφαλείας μα. Θα πρέπει ε, να βρεθεί τρόπος να βελτιωθούν αυτές οι δομέ. Δεν ξέρω αν χρειάζονται και επενδύσει είναι απλώς θέμα οργανωτικό. Είμαι βέβαιος λοιπόν ότι θα συνεργαστούμε καλά και σε επικοδομητικό πνεύμα με τις τροπολογίες θα βελτιώσουμε την έκθεση και μπορούμε θα πρέπει να δούμε και τα θέματα της Γενικής Γραμματείας του Κοινοβουλίου και θέματα επικοινωνίας. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Ο κύριος Μπόκρος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η επιστολή του Επιτρόπου Γιάννου Λεβαντόφσκη είναι ένα πολύ σημαντικό κείμενο. Και το πνεύμα του κειμένου ξεπερνάει κατά πολύ το γράμμα του κειμένου. Διότι το κείμενο ουσιαστικά αναφέρεται στην πρόθεση της Κομισιόν πώς θα κάνει τις δικές της προτάσεις για τον προπολογισμό. Αλλά παρουσιάζει νομίζω σωστά την ε, θέση της Κομισιόν στη σύνολό και μας δίνει μια πρόγευση της συμπεριφοράς και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το να βλέπουμε λοιπόν αύξηση 4% φαίνεται να είναι τελείως εξωπραγματικό για, αυτή τη χρονιά. Όσοι είναι αισιόδοξοι για την οικονομική ανάπτυξη στην Ένωση, έχω να τους πω ότι η κρίση συνεχίζεται και ακόμα είμαστε στη μέση της κρίσης. Το ίδιο ισχύει για την Ισπανία και την Πορτογαλία. Ας λάβουμε λοιπόν υπόψη μας ότι ο ευρωπαϊκός προπολογισμός πρέπει να είναι πολύ λιτός και θα είναι όσο και να θέλουμε να τον μεγαλώσουμε εμείς. Και είναι σημαντικό αυτό που είπε, που είπαμε πολύ και η συγγήτρια ότι δηλαδή αν θέλουμε να έχουμε έναν προϋπολογισμό με ισχυρές προτεραιότητες πρέπει να επιλέξουμε και αρνητικές προτεραιότητες. Και προειδοποιώ κατά κάποιο από την εισηγήτρια μην παρατονίζει πολύ τις συνέργειες με τον προπολογισμό της Ένωσης και των εθνικών προπολογισμών διότι αυτοί οι προπολογισμοί έχουν τελείως διαφορετική διάρθρωση. Οι εθνικοί προπολογισμοί στο 90% αναφέρονται σε τρέχουσες δαπάνες. Να, εσείς, και το είπατε εσείς, αυτό που θέλετε να πετύχετε, ο προπολογισμό της Ένωσης να βοηθάει την οικονομική ανάπτυξη, που σημαίνει ότι δεν είναι ένας προπολογισμό που στηρίζεται στις πάγιες δαπάνες θα πρέπει να στηρίζεται περισσότερο σε επενδύσεις. Και στο σημείο αυτό συμφωνώ με την Helga Trippel, διότι αυτό ακριβώ είναι το ζητούμενο. Αν θέλουμε οικονομική ανάπτυξη, πρέπει να δίνουμε περισσότερα λεφτά για επενδύσεις. Και στους ανθρώπους, στην έρευνα, κινητικότητα των νέων, εκπαίδευση, κατάρτιση, και όπου υπάρχουν πραγματικά συνέργειες όπως η υποδομή μεταφορών και ενέργειας αλλά τι να κάνουμε πρέπει να πούμε και την πικρή αλήθεια το Ταμείο ε, της ε, globalization όπως το λέμε αυτό ας το αφήσουμε γιατί είναι ένας τρόπος ε, για τρέχουσες δαπάνες που θα προφυλάξουν το status quo ουσιαστικά. Το ίδιο ισχύει και για το κείμενο του συναδέλφου Φερνάντες. Θεωρώ ότι αν δεχτούμε το μήνυμα της Επιτροπής Λεβαντόφσκη πρέπει και εμείς να κάνουμε την ίδια εξοικονόμηση πόρων κοδηλίων στον προπολογισμό μας που σημαίνει περικοπές ίσως και το σπίτι του ευρωπαϊκού πολιτισμού κλπ. Για να έχουμε ένα, ένα περιθώριο για το μέλλον, αν και όπως ξέρουμε μέχρι τότε μπορεί να μην είμαστε πια παρόντες. Χρειαζόμαστε λοιπόν να ορίσουμε σωστά τις προπατεραιότητες μας και θετικά και αρνητικά διότι αυτός ο προπολογισμό τελείως διαφορετικός από τους εθνικούς προπολογισμού, πρέπει να είμαστε υπέρ των ε, επιμέρους ε, κονδυλίων και χρηματοδοτήσεων συμπεριλαμβανομένων και των επενδύσεων. Πρόεδρε, ευχαριστούμε. Μας έφερε εδώ το, το, το Γιάννος με το πνεύμα του κατά κάποιο τρόπο να πλανάται με στην αίθουσα κρατώντας ένα μεγάλο ψαλίδι στο χέρι. Κυρία Μπέρμαν. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ σύντομα ήθελα εγώ το λόγο για το θέμα των αποκεντρωμένων οργανισμών, agencies, που αναφέρονται στη σελίδα 8 στην έκθεση κυρίας Μπασάν. Νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι οι οργανισμοί αυτοί είναι ε, βασικά ένα θέμα κύρους των διαφόρων κρατών μελών. Εγώ δεν είμαι καθόλου εκείνη που θα αμφισβητήσει την αποτελεσματικότητα, τη σκοπιμότητά του. Δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι του χρειαζόμαστε απαραίτητο στου οργανισμού, Έχουν τη χρησιμότητά του. Θα ήθελα να τονίσω όμω το εξή και να προτείνω ε, για την εξοικονόμηση πόρων να κάνουμε μία έρευνα ε, της λειτουργίας τους ε, μήπως υπάρχει δυνατότητα σε κάποιους από τους οργανισμούς αυτούς να εξοικονομηθούν ε, πόροι λειτουργικοί. Ευχαριστώ. θα το θέσουμε υπόψη της Γιούτα Χάουκ που χρειάστηκε να βγει. Ε, κύριος Γκοντμάνης, ε, σύντομα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να είμαστε επαναστάτες ιδιαίτερα. Αν πάρουμε το έγγραφο εργασίας που λέει σχέδιο προπολογισμό για το 2012. Βλέπουμε τις διαφορές στα ποσοστά και τα νούμερα. Και αυτό που άκουσα είναι ότι το Συμβούλιο θα είναι πιο σκληρό, πιο συντηρητικό, μάλιστα. Αν όμως, αν θέλουμε ε, να έχουμε για μας μια αφετηρία, μια βάση, δεν θα μπορούσαμε να πούμε το ίδιο ποσοστό, το ίδιο, ε, ποσοστό πληρωμών όπως είχαμε την προηγούμενη χρονιά, 2,9%, όχι παραπάνω. Είναι ρεαλιστικό αυτό ή όχι. Θα δούμε τις τελευταίες προβλέψεις της Ένωσης του Φθινοπόρου. Τελευταίες προβλέψεις είναι αυτές. Της Κομισιόν. Βλέπουμε αύξηση του ΑΕΠ φθινόπλου 2010, άνοιξη 2010 για όλη την Ευρώπη. είναι 1,7%. Δηλαδή το ίδιο. Το 2010 ήταν διαφορετικά στο μισό. Στο 1 ήταν 0,8% και το φθινόπωρο και την άνοιξη ήταν 1%. Αν δείτε όμως την πρόβληψη του 2012 με βάση την Κομισιόν, αύξηση 2% και η κύρια διαφορά είναι στις επενδύσεις. Το φθινόπωρο οι προβλέψεις, οι επενδύσεις προβλεπόταν 2,4%, διπλάσιο δηλαδή από ό,τι είχε προγραμματιστεί την Άνοιξη. Δηλαδή ουσιαστικά η Κομισιόν θεωρεί ότι το τμήμα του ΑΕΠ που είναι για επενδύσεις θα αυξηθεί πολύ τρεις φορές παραπάνω Μπορούμε να το πάρουμε αυτό σε βάση για να πούμε στο Συμβούλιο. Αυτό είναι ένα σχέδιο προεπολογισμού αν το συγχρηματοδοτήσουμε αυτές τις επενδύσεις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μόχλευση σε σχέση με τις εθνικές επενδύσεις. Γι' αυτό θεωρώ ότι αν ξεκινήσουμε με ένα όριο, βέβαια θα εξαρτηθεί από αυτό που μας έστειλε ως υλικό η Κομισιόν, την πιο συντηρητικό, να πούμε να είναι το ίδιο ποσοστό που είχαμε μεταξύ του 10-11. Είναι δυνατόν, βλέποντας τα νούμερα της αύξησης του έπνα, να προστατεύσουμε κάπως το σημείο αυτό. Και μετά, στη συνοχή και τη γεωργία. Στη συνοχή μεν είναι σαφές ότι είναι δυνατόν να υπολογίσουμε πόσα λεφτά χρειαζόμαστε αν δεν έχουμε σημαντική αύξηση της ταχύτητας απορρόφησης. Δύο φορές πιο πάνω από ό,τι είχαμε προγραμματίσει το 2011. Αν η αύξηση είναι 10 11% όπως ήταν στο παρελθόν, τότε ίσως τα χρήματα να μην είναι 0,4% να μπορεί να είναι λιγότερα. μερικές σκέψεις όχι πολύ κλασικές, κάπως επαναστατικές θα έλεγα, πρόεδρος. Αγαπητέ συνάδελφοι, πράγματι η οικονομική ανάλυση είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Μία δυσκολία μας είναι το πρόβλημα πιστώσεις υποχρεώσεων και πληρωμών. Γιατί οι πιστώσεις πληρωμών είναι περίπου όσο και υποχρεωτικέ δαπάνε. Καταργήσαμε τη διάκριση μεταξύ υποχρεωτικών και μη υποχρεωτικών δαπανών στον κοινοτικό προπολογισμό με τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Νομικά όμω, όταν αναλαμβάνουμε μια υποχρέωση και έγινε η δουλειά, προσλήφθηκε κάποιο, α πούμε, βάσει μια υποχρέωση, πρέπει να πληρωθεί μετά. Τη δουλειά αυτή που έγινε, ο, ο ο οποίο προσλήφθηκε. Η μεγάλη δυσκολία για φέτο είναι ότι είναι αδύνατο να μην αυξήσουμε τα κονδύλια πληρωμών. Και το τεράστιο λάθος που διαπράχτηκε από τις κυβερνήσεις ήταν να δευματευθούν τις πιστώσεις πληρωμών. Ενώ πολιτικά το σημαντικό και οικονομικά αυτό που είναι σημαντικό ως χρηματοδότηση είναι οι πιστώσεις υποχρεώσεων. Μπορεί να μπλοκάρεις τις πιστώσεις αυτές ή να τις μειώσεις οι πιστώσεις πληρωμών εξαρτώνται από ποσά τα οποία δεσμεύθηκαν την προηγούμενη χρονιά και πίσω. Ευχαριστώ όλους τους που μίλησαν. Οι εισηγητές θα τους δώσω το λόγο για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Δύο-τρεις σκέψεις μόνο. Η εισηγήτριά μας κυρία Μπαλζάνη προτείνει δύο κείμενα πολιτικά. Το ένα είναι ένα έγγραφο εργασίας για βάση συζήτηση με τις εξειδικευμένες επιτροπές του Κοινοβουλίου και το δεύτερο είναι ένα σχέδιο ψηφίσματος για την Ολομέλεια σύντομο σαφές, συγκεκριμένο έτσι ώστε η Κομισιόν όπως σωστά ζήτησε ο Επίτροπος Λεβαντόφσκι, όταν θα ετοιμάσει το σχέδιο προπολογισμού, να μην βρεθεί σε μια κατάσταση όπου μόνο ο ένας, το ένα σκέλος της αρχής του προπολογισμού θα έχει πει ναι και το άλλο ακόμα να μην έχει πάρει θέση σε επίπεδο, ανώτατο επίπεδο λέει ολομέλεια. Όσον αφορά το Συμβούλιο, το Συμβούλιο ήδη ενέκρινε τις κατευθυντήριες γραμμές και με βάση την παράδοση ήθεστε το Συμβούλιο έτσι το ζούμε και έτσι το αγαπάμε θα έλεγα. Τώρα για τις αρνητικές προτεραιότητες. Διαπιστώνω ότι κάθε χρόνο κυκλοφορεί αυτή η ιδέα. Και εγώ ίδιος το ζήτησα στο παρελθόν. Και κάθε χρόνο την παίρνουμε πίσω γιατί πολιτικά είναι πολύ δύσκολο. Κατά γνώμη μου, το λέω για τους συζητητές να το σκεφτούν. Υπάρχουν δύο τρόποι να προτείνουμε αρνητικές προτεραιότητες, δηλαδή ουσιαστικά μείωση κονδυλίων σε ορισμένε γραμμές. Ο ένας τρόπος είναι εμείς, Επιτροπή Προπολογισμού, να μην ακούσουμε τις άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Ξέρουμε πώς μπορούμε να κάνουμε τις αρνητικές προτεραιότητες. Αλλά αν ακούσουμε την Επιτροπή Γεωργίας, την Περιφερειακή, την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, στην οποία δεν αρνούμαστε ποτέ τίποτα, ξαφανίζονται οι αρνητικές προτεραιότητες. Ο Πιέρ είναι εδώ και η Ουγγρική Προεδρία και τον χαιρετίζω και τον ευχαριστώ για την κατανόηση που επέδειξε πέρυσι ε, εξ ονόματος της Βελικής Προεδρίας. Το σύστημα των Υπουργών Οικονομικών στην Ένωση δουλεύει χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους άλλους υπουργούς που δαπανούν και κάνει ό,τι θέλει. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεύτερη μέθοδος να βρούμε μια αντικειμενική βάση, ας πούμε, τις γραμμές όπου δεν δαπανήθηκαν ή τουλάχιστον επαρκώς τα κονδύλια στο παρελθόν. Πολλοί από εσάς το προτείνατε αυτό. Με αυτό πρέπει να αρχίσουμε. Δυστυχώς όμως η εμπειρία μας δείχνει ότι συνήθως η πιο ενδιαφέρουσα πολιτική, η πιο καινοτόμα πολιτική και η πιο δύσκολη είναι αυτή που στην αρχή καθυστερεί. Δεν ξέρω αν ε, η εισηγήτρια θα να, ή ο εισηγητή θέλει να προσθέσετε κάτι. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Σύντομα, παρακαλώ. Αρχίζουμε τον κύριο Φερνάντε. Ευχαριστώ πολύ, ε, κύριε Πρόεδρε. Θα πω κάτι που είπα και την περασμένη φορά. Θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι θεσμικά όργανα που λειτουργούν με καλή πρόθεση, καλοπροαίρετα και αναλαμβάνουμε ευθύνες και υποχρεώσεις που θα πρέπει να τιμούμε. Αυτό το θέμα του οίκου της ευρωπαϊκής ιστορίας ήταν μια ε, υπόθεση που αναλάβαμε στο παρελθόν και το μόνο τώρα που θα πρέπει να συζητούμε είναι πώς θα ανταποκριθούμε σε αυτή την ανάληψη υποχρέωση. όχι πώς θα την καταργήσουμε. για τους βοηθούς το ίδιο ισχύει. Είπαμε ότι εάν τηρηθούν κάποιες προϋποθέσεις θα λυθεί το θέμα αυτό των ε, βοηθών μας. Τώρα, ως προς την έκθεση και πού βρισκόμαστε. Αυτή τη στιγμή συζητούμε τις πολιτικές προτεραιότητες και θα εγκρίνουμε δύο ψηφίσματα. Το ένα για τις πολιτικές προτεραιότητες και το άλλο για την κατάσταση προβλέψεων. Μα δεν μιλάμε ακόμα καν για κατάσταση προβλέψεων. Αυτές οι προβλέψεις θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις δικές μας πολιτικές προτεραιότητες αυτό είναι η κατάσταση προβλέψεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο είναι διαφορετικά όργανα. Είναι και πολιτικά όργανα, δεν είναι μόνο ε, εκτελεστικά. Ελπίζω να συμφωνήσουμε. Τώρα, τι θα γίνει με την επιστολή του Επιτρόπου κ. Λεβαντόφσκη. Στις του μηνό κατέθεσα εγώ την έκθεσή μου και η επιστολή φέρει επίση ημερομηνία 3 Φεβρουαρίου. Δεν μπόρεσα. Δεν ήταν δυνατό να συμπεριλάβω το κείμενο της επιστολής στην έκθεσή μου, διότι δεν είχαμε λάβει γνώση ακόμα ε, του περιεχομένου της. σε ό,τι αφορά το προπολογισμό από μηδενική βάση, τις μη πάγιες δαπάνε και την κτηριακή πολιτική του Κοινοβουλίου, εγώ περιορίστηκα στο να χρησιμοποιήσω κάποιες έννοιες ε, που με απασχολούν και εμένα και την πολιτική μου ομάδα και ελπίζω να συμφωνούν και άλλες πολιτικές ομάδες. Το ίδιο ισχύει και για τις πάγιες και μη δαπάνεση, η πολιτική αποτελεσμάτων, η πολιτική που να βασίζεται στις επιδόσεις μας. Αυτό δεν εφαρμόζεται σε όλες τις πολιτικές, αλλά στην πολιτική επικοινωνίας γίνεται αυτό ή στην κτηριακή πολιτική που έχει συζητηθεί επανειλημμένα. Και και μελέτη. Εμείς θέλουμε μια πολιτική ε, μεγάλης εμβέλειας. Τι σημαίνει τώρα εξυγίανση των προϋπολογισμών. ότι από το 2012 και το 13 ε, θα πρέπει να επέλθει μια σταθερότητα στον προϋπολογισμό. Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν ένα προϋπολογισμό χωρίς εκπλήξεις. Βέβαια, από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην κατηγορία 5. Τι θα γίνει με τον προγραμματισμό από εκεί και πέρα για την επόμενη περίοδο και πόσο σταθερό θα είναι ο προπολογισμό με βάση τις περικοπές και τις οικονομίες που θα γίνουν. Ελπίζω να μας κάνει προτάσεις στο Προεδρείο για να απαντήσει στις προτεραιότητες ε, που έχουμε. Και σίγουρα, για να απαντήσω στον κύριο Άλβαρο, μπορεί να χρειάζονται περισσότερα χρήματα, δεν είναι μόνο ποσοτικό το θέμα, χρειάζεται και καλύτερη λειτουργία. Είμαι βέβαιος ότι το Προεδρείο θα μας κάνει τις προτάσεις του ε, σχετικά. Δεν μπορούμε όμως να λησμονούμε το στόχο μας η αριστεία παραμένει και η αριστεία στην νομοθετική λειτουργία, γιατί αυτό το απαιτούν από εμά οι πολίτες και θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να νομοθετούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και επαναλαμβάνω ότι ο προπολογισμό του 12 και του 13 θα αποτελέσει αναφορά για του επόμενου προπολογισμού του ε, πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου. Σα ευχαριστώ για τα σχόλιά σα. Είμαι απολύτω στη διάθεσή σα για να συνεργαστούμε, για να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την έκθεση και τα ποσά. Πάντως προς το παρόν ε, μιλούμε για τις πολιτικές προτεραιότητες. Για ποσά όχι ακόμα. Ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Φραντζέσκα παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα απαντήσω στις συναδέλφους που ανάφεραν τις προτεραιότητες και ξεκινάω την πρόταση ψηφίσματος που θα την παρουσιάσω στις 3 Μαρτίου. Η προσπάθειά μας μετά αυτό που έγιναν πέρυσι και την ε, έντονη θέση που πήραμε σε πολλές συζητήσεις και τον Ιούνιο για την οικονομική διακυβέρνηση και το ψήφισμα του Δεκεμβρίου επίσης και το σημαντικό πακέτο της, 20, της 9ης Σεπτεμβρίου σημαντικό στην ιστορία της Ένωσης από αυτά βγαίνει ένα σαφές μήνυμα η Ευρώπη έχει μια στρατηγική δεκαετίας και χρειάζονται προσπάθεια, προσπάθειας σύγκλησης γιατί τα χρήματα δεν είναι επαρκή, θα πρέπει να δημιουργηθεί κρίσιμη μάζα έτσι και να αποφευθεί ο περισπασμός και η διάσπαση. Ξεκινάει και το ευρωπαϊκό εξάμεινο και γι' αυτό η πρότασή μου είναι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, το μεγάλο στίγμα θετικό με την έννοια αυτή της Ένωσης, να είναι ένα εργαλείο και ένα μήνυμα και για τους εθνικούς προπολογισμού. Άρα, προτεραιότητα για μας πολιτικά και θεσμικά και για λόγους μη ανακολουθίας σε σχέση με αυτά που ήδη αποφασίσαμε θα πρέπει να, όλα αυτά να κινούνται μέσα στο πλαίσιο της στρατηγικής 2020. Έχουμε την ετήσια έκθεση της Κομισιόν για την Οικονομική Ανάπτυξη που τονίζει τις προσπάθειες που χρειάζονται για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Η στρατηγική του 2020 είναι πέντε συγκεκριμένοι χρήσιμοι στόχοι ε, πολέμηση αλλαγής του κλίματος, ε, ε μη κοινωνικό αποκλεισμό, δημιουργία θέσεων απασχόληση, έρευνα κλπ. Η πρόταση λοιπόν είναι να επικεντρώσουμε την ενέργεια και τους προπολογισμού με βάση αυτά που αποφασίσαμε και αποφάσισαν και οι Κομισιόν και εμείς εγκρίναμε το Δεκέμβριο για τα μεγάλα θέματα της Ευρώπης 2020 για να αποφύγουμε κι άλλου είδους ήτες γιατί η, το πρόβλημα με τη Λισαβόνα ήταν ότι υπήρξε δυσκολία στο να δημιουργηθεί αυτή η κρίσιμη μάζα. Το δικό μου λοιπόν ψήφισμα που θα σας το παρουσιάσω στις 3 Μαρτίου θα είναι μια σαφής πρόταση και περιγραφή της στρατηγικής μας και ότι μένουμε μέσω σε αυτό το πλαίσιο προτεραιοτήτων της Ένωσης για την επόμενη δεκαετία. Αρνητικές προτεραιότητες. Πρέπει να γίνουν και εδώ προτάσεις. Σε θετική κατεύθυνση, δηλαδή αρνητικές προτεραιότητες, δεν είναι αυτά όλα που αποδείχθηκαν λάθος ή που δεν απέδωσαν. Μερικές φορές οι προτεραιότητες γίνονται αρνητικές γιατί δεν συμφωνούν ε, με την χρονική συγκυρία, παραδείγματος χάρη. Άρα χρειάζονται νέες θετικές προτεραιότητες. Είναι και αυτές ένα εργαλείο πολιτικής ευελιξίας του προπολογισμού. Να αλλάξουμε τις προτεραιότητές μας είναι ένας τρόπος να προσαρμόσουμε τον προπολογισμό στους καιρούς. Αυτό το κάναμε όταν αρχίσαμε να συζητάμε τη διάρκεια των δημοσιονομικών προοπτικών. Ας γίνουν λοιπόν και εδώ προτάσεις Συγκεκριμένε, Θα είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό για τις άλλες επιτροπές και να το ζήσουμε σαν ένα εργαλείο που θα μας οδηγήσει σε νέες προτεραιότητες μια ακόμα μορφή και διάσταση ευελιξίας του προπολογισμού. Χρήσιμη μέσα στην περίοδο των οικονομικά ισχυνών αγελάδων που διανύουμε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ Φρανσέσκα. Στις προσεχείς ημέρες η Φρανσέσκα θα έρθει σε συνεννόηση με τις ε, υπηρεσίες του Κοινοβουλίου και για τις 23 Μαρτίου θα μας υποβάλει ένα έγγραφο για τις γενικές προτεραιότητες και τη στρατηγική ενόψη της ψηφοφορίας στις 16 ε, Μαρτίου στην Επιτροπή και την, την έγκριση Ολομέλεια την 1η του Απριλίου. Και βεβαίως έχουμε την, ε, τον, προγραμματισμό για έγκριση του σχεδίου στις 20 Απριλίου, στο σύνολο του επιπλήξμου. Αγαπητοί φίλοι, έχουμε πολλά θέματα να συστήσουμε, πολύ λίγο χρόνο, θα προχωρήσουμε στο δυνατόν πιο γρήγορα. Αυτά τα οποία έχουμε μέχρι τώρα όμως ε, συζητήσει, πιστεύω ότι αξίζαν τον κόπο να αφιερώσουμε λίγο παραπάνω χρόνο. Τα είδαμε και στην ε, περίπτωση της αναθεώρησης συνθήκης με τους συνεχισηγητές πόσο σημαντικά είναι αυτά. Λοιπόν, θα έλεγα πολύ γρήγορα να πάμε στα σημεία 6 και 7, όπου έχουμε να κάνουμε με την ε, κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης, ύστερα από τις πλημμύρες, που έλαβαν δυστυχώς χώρα στην Πολωνία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, την Δημοκρατία της Τσεχίας, την Κροατία και τη Ρουμανία. Επί της ουσίας, αρμόδιος ηγητής είναι ο κύριος Μπέγκε. Για τον διορθωτικό προϋπολογισμό αρμόδια είναι η Συντόνια από ό,τι όμως φαίνεται, το Συμβούλιο δεν είναι σε θέση να λάβει απόφαση. Θα προτείνω λοιπόν στον Ράινερ να μας ε, περιγράψει πολύ γρήγορα την πρόταση και να ε, αναβάλουμε τη λήψη αποφάσεως μέχρι ότου το Συμβούλιο έχει ε, προσδορίσει θέση του. Ράιμερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε πάρα πολύ σύντομα. Ήδη σε προηγούμενη συνεδρίαση είχαμε συστήσει τα θέματα των ε, αριθμητικών στοιχείων ως προς την ε, κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης ε, για την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, την Τσεχία, την Ρουμανία. Και βέβαια επιπλέον την υποψήφια για ένταξη Κροατία. 182 εκατομμύρια. Συνολικά τα έγγραφα έχουν την κατανομή, τη λεπτομερέστερη κατανομή. Ύστερα από την ολοκλήρωση μιας ε, επόδυνη διαδικασίας του προϋπολογισμού, καταλαβαίνετε ότι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και περιέργεια περιμένουμε να δούμε πώς θα χειριστεί το θέμα αυτό η Συντόνια για το πρόσθετο, για το δορθωτικό προπολογισμό ενώ κινητοποίηση του Ταμείου Ελεγγύης. Εγώ νομίζω ότι θα ήταν καλό να περιμένουμε και τη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Επιτροπής η οποία δυνάμει της εσωτερικής μας διαδικασίας ε, πρόκειται να τοποθετηθεί και θα έλεγα την στην επόμενη μας συνεδρίαση, στην Επιτροπή των Προπολογισμών, να ε, προχωρήσουμε, εφόσον η κατάσταση είναι όρημη, σε λήψη αποφάσεως. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Η Συντόνια θέλει να πει δύο λόγια. Λεφτά μπορεί να μην έχει να δώσει, αλλά θα πει την κουβέντα της. Πρόεδρε, το πιο σημαντικό θέμα νομίζω είναι να εξηγήσει το Συμβούλιο που διαπιστώνει εμπόδια, που βλέπει τα προσκόμματα στη λήψη αποφάσεως. Τι το εμποδίζει να λάβει την απόφαση. Και επίσης θα ήθελα να συμφωνήσω με τον κύριο Μπέγκε ότι πρέπει να διατεθούν τα κονδύλια αυτά. Εγώ έχω την ε, ε, πρόταση, όπως είπα, για το διορθωτικό προϋπολογισμό και όπως είπα και νωρίτερα πρέπει η ανταπόκριση, η αντίδραση σε, εθνικές, σε φυσικές καταστροφές ε, με κινητοποίηση του Ταμείου Ελεγγύης να είναι ταχύτατη. Δεν βλέπω γιατί θα πρέπει να καθυστερήσουμε, γιατί θα πρέπει να καθυστερήσει αυτή η διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χάρτον, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω την συγκήτρια πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτόματα το πληρώνει αυτό, είναι ευθύνη των κρατών μελών, γιατί είχαμε ήδη κάποιες επαφές με ε, κάποιους Ούγγρους και από ό,τι φαίνεται έχουν χτιστεί πάρα πολλά σπίτια σε ε, περιοχές που ε, πλημμυρίζουν και που δεν τις ασφαλίζουν καν ασφαλιστικές εταιρείες γιατί η κυβέρνηση ίδια λέει ότι δεν μπορούν εκεί να χτίζουν σπίτια, είναι τόσο μεγάλος ο κίνδυνος πλημμυρών. Οπότε τι εμείς πάμε και πληρώνουμε αυτομάτως αποζημιώσεις, δεν είναι ευθύνη των κρατών μελών αυτό. Oui, Sidonia. E, Πρόεδρε, άκουσα με ενδιαφέρον την παρέμβαση του συναδέλφου. Λίγες είναι οι χώρες πλην της δικής σας που έχουν τόσο πολλά κτίρια ανεγύρι σε περιοχές που παρουσιάζουν το φυσικό φαινόμενο της πλημμύρας σε ορισμένε περιόδους. Θα πρέπει βεβαίως να δούμε τι είδους απώλειες υπάρχουν, τι είδους απώλειες σε υποδομές και πώς μπορούν να αποκατασταθούν αυτές με προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει ουδεμία μορφή ασφάλισης. Η ιδιωτική, η ιδιωτική ε, περιουσία Φερρυπίνη αποκλείεται από το Ταμείο Αλληλεγγύης. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ένα αναμονή μιας απόφασης του Συμβουλίου. Αφήνουμε το θέμα αυτό και προτείνω να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα με την Ίγκε Γκρέσλε, η οποία συμφωνεί στο σημείο 10 γιατί και εκείνη χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο για να ετοιμάσει ένα γραφείο εργασία. Αναβάλλεται λοιπόν το σημείο 10. Κυρία Γκρέσλε, μέρα τη μέρα και ε, τα Σαββατοκύριακά τη ακόμα το υπογραμμίζω. Συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή και το Συμβούλιο και είμαι βέβαιος ότι το έγγραφο το οποίο θα μας υποβάλει θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αφήνουμε λοιπόν το σημείο 10 και περνούμε στο σημείο 11, πρόγραμμα στήριξης της περαιτέρω ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης θαλάσσης πολιτικής με τον κύριο Ντομινίκ Ρικέ. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ενθυμίσω ότι πρόκειται για ένα έγγραφο που αναφέρεται σε μια πολιτική ε, σχετική με το 40% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη έχουν υπογραμμιστεί η σημασία αυτής της πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι προπαρασκευαστικές δράσεις, τα πιλωτικά σχέδια ολοκληρώνονται, κλείνουν δηλαδή μέσα στο 2011 και θα πρέπει να προσβληθεί για την συνέχεια αυτών των, εργα... των δράσεων και των σχεδίων ε, ένα πλαίσιο. Προτείνονται λοιπόν δύο νέες γραμμές στον προπολογισμό στον τίτλο 11 του προϋπολογισμού, στο δεύτερο τμήμα, χρηματοδότηση τριετή από το 11 έως το 13 για 50 εκατομμύρια στη, στο, από το δημοσιονομικό περιθώριο του τίτλου 2. Προτείνεται να αντιληφθούν τα κονδύλια αυτά και προτείνω να ακολουθήσουμε την Επιτροπή στις προπαρασκευαστικές αυτές δράσεις και τα πιλωτικά σχέδια ολοκληρωμένης της πολιτικής για τις θάλασσες με αυτά τα 50 εκατομμύρια λοιπόν για τρία χρόνια στο τμήμα υπαριθμών 2, αυτό το υπογραμμίζουμε στην έκθεση και βεβαίως και στο νομοθετικό σχέδιο. Τροπολογίες. Έχουμε καταθέσει μόνο για να ε, ξεσφαλίσουμε ότι δεν θα επιδοτηθούν αυτές οι ε, προκηρύξεις για εκδήλωση ενδιαφέροντος κατανομή συγκεκριμένη με κριτήρια συγχρηματοδότησης, κατανομή σε τίτλους, έκθεση μέσω πρόθεσμη της εκτέλεσης των προγραμμάτων, των σχεδίων και συμμετοχή του Κοινοβουλίου στις διαδικασίες ε, έγκρισης του ετήσιου προγράμματος και της αναθεώρησής του. Και στο νομοθετικό τμήμα αναφέρονται συγκεκριμένα οι ε, τίτλοι οι γραμμές του προϋπολογισμού δηλαδή. Αυτά ήταν όλα. Απλώς επιβεβαιώνουμε τη βούλησή μας να στηρίξουμε την πρόσθεση επιτροπή για τα 5 εκατομμύρια. Α, τα αντλούμε αυτά τα ποσά από το περιθώριο του τμήματος 2 και εισάγουμε, αυτό είναι που προτείνω εγώ ως βελτίωση, επιπλέον ελέγχους στην εφαρμογή και στην αποδοτικότητα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Γκρελιέ. Δεν σας δώσω το λόγο ακόμα. Κυρία Γκρίλια, ναι, ναι, όπως είπατε. Ε, Δύο-τρία σημεία μόνο και μια ερώτηση. Είπε ο εισηγητή μα ότι χρηματοδοτείται αυτή η πολιτική από πιλωτικά σχέδια και προπαρασκευαστικέ δράσει και σε αυτό το στάδιο μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η υπηκοδότηση με 50 εκατομμύρια αποτελεί μια μικρή έστω πρόοδο. Πλην όμως ε, στην προοπτική των πολύ σημαντικών κοινοτικών προκλήσεων που παρουσιάζει το θέμα αυτό, η θεματολογία αυτή, νομίζω ότι θα ήταν καλό να υπογραμμίσουμε στην έκθεση την αναγκαιότητα για δημιουργία νομική βάση, νομικών βάσεων, ολοκληρωμένη πολιτική για τι θάλασσε, που να αξίζει, για τις θάλασσες, που να αξίζει αυτό τον τίτλο, και βεβαίω να έχουμε και μια συζήτηση διεξοδικότερη για τι δημοσιονομικέ προοπτικέ. Και είμαι ότι ήδη είναι πεπισμένο γι' αυτό η δεν χρειάζεται να και θα ήθελα επίση να ε, επισημάνω ότι θα πρέπει το Συμβούλιο να κάνει προσπάθεια συνοχή στην υπόθεση αυτή, γιατί αν δεν υπάρχει κοινοτική πολιτική, ε, βλέπουμε αντίστοιχα ότι χαλαρώνει και η σχετική ε, σημασία που αποδίδεται σε εθνικό επίπεδο. Βλέπουμε ότι οι Βρετανοί επί παραδείγματι έχουν εγκαταλείψει την υπόθεση ε, της ε, ρημούλκησης μεγάλων πλοίων στα στενά της Μάνχης και μάλιστα σε, πίνοντας ένα ποτηράκι μου είπαν ανεπίσημα ότι επειδή είναι αντίθετοι οι άνεμοι δεν τους βολεύει αυτή η δουλειά και την έχουν αφήσει στην πρωτοβουλία των Γάλλων. Δεν τους συμφέρει δηλαδή. Αυτά για να προχωρήσω λοιπόν, ε, ναι, βλέπω σε ποιο σημείο ε, προβλέπετε την άντληση των ποσών, αλλά πώς ακριβώς και δεύτερον η κατανομή των στόχων, των ποσών στόχο, πώς μπορεί να γίνει. Θα μου ευγνώμων αγαπητέ Ντομινίκ να μου έδινε απαντήσεις. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος και ευχαριστώ πολύ για το είπατε για τους ανέμους στη μάχη. Χωρίς να είμαι ναυτικός, οι Ισπανοί φίλοι εδώ θα θυμούνται ίσως ότι η ανίκητη ναι. αρμάδα του βασιλείου της Ισπανίας απέτυχε ακριβώς σε μια απόπειρα να καταλάβει τα βρετανικά, τις βρετανικές νήσους χάρη στον Φράνσις ε, Drake, ε, Blake και ε, τους Drake και τους θαραλέους ε, ε ναυάρχους του Βρετανικού στόλου αλλά και χάρη στα καπρίτσια του Ποσειδώνα. Παρακαλώ για την απάντηση ο κύριος Ρικέ. Ναι, ευχαριστώ για τα περιθώρια όπως είπα, από εκεί θα αντιληφθούν τα ποσά και όπως είπα ε, προτείνεται και μια νομοθετική διατύπωση με δημιουργία ουσιαστική αυτού του περιθωρίου, δηλαδή θεσμική δουλειά θα εγγραφεί ουσιαστικά μέσα στο προπολογισμό αυτό το σύνολο των ε, σχεδίων και προπαρασκευαστικών πράξεων. Και όπως είπα, ναι, ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει αυτή τη δουλειά, αλλά ζητούμε και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να επανέρχεται κάθε χρόνο και να προσδιορίζει έστω και τις, λεπτομέ... και τις λεπτομέρειες μάλλον των σχεδίων σε κάποια συγκεκριμένα σημεία. Δεν θέλαμε δηλαδή να δώσουμε απλώς 50 εκατομμύρια μέσα σε ένα πλαίσιο χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένα υπομέτρα. Θέλουμε να έχουμε μια σαφή επισκόπηση κατάστασης. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος προθεσμία για τις τροπολογίες 18 Φεβρουαρίου στις 10. Είχαμε πει ότι ίσως να το επαναφέραμε για τη συνεδρία στις 3 Μαρτίου το θέμα αυτό, αλλά αν δεν χρειαστεί θα το αφήσουμε. Ψηφοφορία προβλέπεται στην συνεδρίαση της Επιτροπής μας 15 και 16 Μαρτίου. Και τώρα προτείνω να περάσουμε στο σημείο 13 με την κυρία Χέρτσοκ ενδιάμεση επισκόπηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων πλοήγησης μέσω δορυφόρου. Αγαπητή κυρία Χέρτσοκ, πολύ γρήγορα. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι στο δυνατόν πιο σύντομη στην υπόθεση αυτή. Προ... Μάλλον έχει καταθέσει μια ενδιάμεση, μια ενδιάμεση μεσοπρόθεσμη επισκόπηση Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς από πλευράς μας δίνουμε την ε, γνωμοδότηση από πλευρά τη Επιτροπή των Προπολογισμών. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ιδιαίτερω ότι. Έχουμε περίπου ακρίβεια 70% με το σύστημα του, ε, το αμερικανικό του GPS και νομίζω ότι έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε σημαντική οικονομία κλίμακο σε ένα τομέα που έχει προβλεφθεί να αυξηθεί στα 150 δισεκατομμύρια ευρώ το 2020, άρα πρόκειται για ένα τομέα που θα έχει μεγάλη ανταγωνιστικότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι το θέμα λοιπόν. Η πρώτη αλλαγή εμφανίστηκε ήδη το 2007. Ήταν ανεπαρκής δηλαδή η χρηματοδότηση για, το, για τα προγράμματα GNSS και έτσι στην ε, αναθεώρηση των ισιουσών τώρα δημοσιονομικών προοπτικών στο, ε, στα 2,4 δισεκατομμύρια για την περίοδο 2007-2013. Μετά το 2007 έγινε το ίδιο και με το Ίτρε. Δηλαδή διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα ως προς τον προγραμματισμό και τη χρηματοδότηση των μακρόπνων σχέδων και επιλογών. Όσο σημαντικές και είναι αυτές. Δεύτερη διαπίστωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ενδιάμεση αυτή επισκόπηση το 2011 δεν προτείνει συμπληρωματική χρηματοδότηση μέχρι το 2013 για την περίοδο που μένει μέχρι το 2013. Λόγω βέβαια αυτού του κόστους, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πολύ σημαντικές καθυστερήσεις προς τις εφαρμογές του προγράμματος GNSS και επιπλέον απώλειες πιθανού ωφέλους. Ένα τρόπος λοιπόν χρηματοδότησης μέσω του 7ου προγράμματος πλαισίου είναι απαράδεκτος ως λύση, εκτός και αν αποφασίσουμε να αναστρέψουμε πρίμναν και να εγκαταλείψουμε την έρευνα και την καινοτομία στο μέλλον. Και δεν νομίζω ότι πρόκειται για μια λύση την οποία σκοπεύει να ακολουθήσει η Επιτροπή μας ή θα έπρεπε να ακολουθήσει. Επίσης, το Γαλιλαίο είναι πρόγραμμα που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρα το δημοσιονομικό μας καθεστώς θα πρέπει να θεσπίσει κατά κάποιο τρόπο ένα σύστημα διαχείρισης και πέραν των κτηρίων της υποδομής που χρειάζεται. Και εδώ πάλι προκύπτουν κάποια ζητήματα. Έτσι, στην ενδιάμεση επισκόπηση του Γαλιλαίου, που είναι πολύ σημαντική ω προ τον προπολογισμό, έχουμε 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ κατεκτήμηση που συλλαμβάνονται σε αυτήν την διάμεση αναθεώρηση για την περίοδο μετά το 2013. Και τα ποσά αυτά θεωρούνται ελάχιστα, ο ελάχιστος προπολογισμό ε, και πρέπει να συμπληρωθεί με 800 εκατομμύρια σε ετήσια βάση. Για το 2014 θα ήθελα να σημειώνω ότι θα έχουμε φτάσει μάλλον σε, ε, στην, στον αριθμό των 18 δορυφόρων, αλλά χρειαζόμαστε συνολικά 28 δορυφόρους για να λειτουργήσει το σύστημα, άρα θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε ε, προχωρήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Άρα λοιπόν εδώ τη ζητούμε για αυτό το δημοσιονομικό έτος και με την έκθεσή μας ε, θα πρέπει να αναζητηθεί το από πού θα χρηματοδοτηθεί αυτό το δημοσιονομικό σχέδιο για το μέλλον. Εάν θέλουμε να περιοριστούμε μόνο στο κοινοτικό προϋπολογισμό θα μπορούσαμε ενδεχομένω να αξιοποιήσουμε το μέσο ευελιξία, όπως είχε με το, ΊΤΡ ή να δεχθούμε ότι ο Ευρωπαϊκό προπολογισμό καλύπτει μέχρι ενό ποσού και η επιπλέον επιβάρυνση, η συμπληρωματικό κόστο καλύπτεται από τα κράτη-μέλη ή από το μέσο για το ίτερ. Δεν θέλω εγώ να το τοποθετηθώ. Εγώ απλώ υποβάλλω την έκθεση. Περιμένω να δω τι θέση έχουν οι σκιώδει συγκητέ. Πιστεύω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτό το σοου, αυτό το σχέδιο. Ανταγωνιστική Ευρώπη δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι μια Ευρώπη η οποία σκοπεύει να θέσει τέρμα σε ένα τέτοιο σχέδιο. Αυτά. Είναι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου. Και περιμένω τις δικές σας θέσεις. Πώς μπορεί να επιταχυνθεί και όχι να διακοπεί ή να ανασταλεί αυτό το πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Είστε σαφέστατος. Ο κύριος Άρτον ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η συγκήτρια λέει θα πρέπει να ανασταλει αυτο το προγραμμα ευχαριστω ειστε ο κυριος αρτον ζητησε το λογο ευχαριστω προεδρε η συγκιτρια λεει θα πρεπει να συνεχιστει το show. Εγώ θα πρέπει να πω όχι the show must go on, the show must stop. Χρόνια ολόκληρα το συζητάμε αυτό το πρόγραμμα. Όλο ρίχνουμε περισσότερα λεφτά. Στο σημείο 5, παραθέτω τι λέει, τονίζει ότι το 1,9 δις που ε, εκτιμάται και μετά το 2013 είναι αμυγός ενδεικτικό και μπορεί να είναι προς τα κάτω εκτίμηση ε, του ποσού που χρειάζεται. Είναι πολλά τα λεφτά, είναι τρομακτικό το ποσό. και παρακαλώ να διαβάσετε στην Επιτροπή την αρμόδια βιομηχανία ότι θα πρέπει να σταματήσει το συντομότερο αυτό το πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Κύριε Ρικέ. Καλά, δεν θέλω να διαφωνήσω με τον κύριο Χάρτον να τον στεναχωρήσω, αλλά εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να συνεχιστεί το πρόγραμμα. Θέλω να κάνω την εξή ερώτηση στην εισηγητρία το Γαλιλαίο και ο Έγνος έχει μια ιδιαιτερότητα. Το διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίδια το πρόγραμμα αυτό. Ε, πάντα γίνεται λόγος για τις δαπάνες. Αυτές είναι επενδύσεις. Ε, στη συνέχεια θα έχουμε και λειτουργικές διαπάνες μετά το 2014, το είπε και η συγκήτρια. Περίπου 800 εκατομμύρια ετησίως για τη διατήρηση του συστήματος. Αλλά κανείς δεν μιλάει για τα έσοδα και θα παρακαλούσα πολύ να μάθω. Έχουμε δημοσιονομική προοπτική όχι για τις δαπάνε αλλά για τα έσοδα και αν ναι, τι θα γίνει, πώς θα τα διαχειριστούν, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζεται το πρόγραμμα επενδύσεων. Εμείς είμαστε μία θηρίδα δαπανών μόνο χωρίς, ε, είμαστε πράκτορες Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο το θέμα αυτό από πλευρά δημοσιονομική στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι υπαρκτό το πρόβλημα και πρακτικό. Ε, κάποια στιγμή θα υπάρχουν έσοδα για τον προπολογισμό. Πώς εγγράφονται αυτά ε, στο δημοσιονομικό πλαίσιο, ε, δεδομένου ότι το διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόγραμμα. Και δεν είναι μόνο πρακτικό το ζήτημα, αλλά και ε, θεωρητικό, έτσι, δημοσιονομικής θεωρίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Ζητήσατε το λόγο εσείς, παρακαλώ, πάρα πολύ σύντομα. πάρα πολύ σύντομα. Δεν ναι, είμαι 100% σίγουρος, λέει ο κύριος Μιλντερ, αλλά θυμάμαι ότι είχαμε κάνει μια συμφωνία ε, για τη χρηματοδότηση του προγράμματος Γαλλία και τότε ήμουν υπέρ και παραμένω υπέρ. Και έλεγε ότι πριν το 2013 Εάν χρειαζόταν επιπλέον χρηματοδότηση, δεν μπορούσε αυτή να επέλθει από τον κοινοτικό προπολογισμό. Κάτι τέτοιο θυμάμαι. Και νομίζω το σημείο 2 ε, δεν είναι ακριβές ότι εκφράζουμε τη λύπη μας διότι η Ευρωπαϊκή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρότεινε τίποτα το νέο. Γιατί νομίζω ότι δεν είναι σε θέση. Βλέπω ορισμένου να ανέβουν καταφατικά, άρα καλά τα θυμάμαι. Ευχαριστώ. Ζητούν και άλλοι το λόγο, λέει ο πρόεδρο, αλλά θα παρακαλούσα να το αφήσουμε εδώ. Όσοι θέλετε ερωτήσει να θέσετε, ελάτε ε, σε επαφή διμερό με την εισηγήτριά μας γιατί δεν προλαβαίνουμε. Ε, θυμίζω την προθεσμία 16 Φεβρουαρίου για κατάθεση τροπολογιών. Έχουμε προβλέψει ψηφοφορία στην Επιτροπή μας 16 και 17 Μαρτίου, έτσι ώστε να γνωμοδοτήσουμε στην Ήτρε, ε, που είναι επί της ουσίας αρμόδια, ε, για τις 31 Μαρτίου. Ευχαριστώ την κυρία Ερτσόκ και τους ομιλητές σας για το 14. Ο εισηγητής κύριος Αλφονσί απουσιάζει. Έχετε όμως λάβει την έκθεσή του, το σχέδιο γνωμοδότησης μάλλον, γιατί γνωμοδοτούμε αρμόδια επί της ουσίας στην Επιτροπή Αλίας. 11 Φεβρουαρίου στις 10 το πρωί λίγη η προθεσμία για τις τροπολογίες για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε στις 3 Μαρτίου. Και ερχόμαστε τώρα στο σημείο 15. Έχουμε δύο μεταφορές πιστώσεων. Η μία φορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι δεν είναι. Δύο διαφορετικές. Στο 15 η Σιδωνία έχετε το λόγο. Αυτή η μεταφορά πιστώσεων αφορά κάποιες ζημίες. Είναι αποζημίωση. Δηλαδή υπάρχει δικαστική απόφαση που διατάσσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταβάλει αποζημίωση 12 εκατομμυρίων ευρώ σε μια εταιρεία ονόματι Sistran είναι μεγάλη ιστορία, παλιά αυτή. Ε, με δύο λόγια θα βρείτε τη σύνοψη, ε, την περιγραφή της μεταφοράς πιστώσεων στο φάκελό σας. Εγώ δεν έμεινα ικανοποιημένη από την ενημέρωση αυτή. Ε, ζήτησα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μου δώσει περισσότερες πληροφορίες, διότι καταρχάς το ποσό είναι τεράστιο, είναι πολλά τα λεφτά, 12 εκατομμύρια ευρώ για αποζημίωση σε μια εταιρεία για παραβίαση των κανόνων περί πνευματικών δικαιωμάτων και copyright και η ίδια η μεταφορά πιστώσεων εδώ είναι 6.300.000 και κάτι ψηλά που είναι επίσης πολλά ε, χρήματα και ως εισηγήτρια είχα την ευκαιρία να δω περισσότερες λεπτομέρειες. Ε, ρώτησα λοιπόν τα εξής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτον, πώς συνέβη τέτοιο πράγμα Δηλαδή η προκήρυξη του διαγωνισμού από το 2003 κατέληξε σε παρεξήγηση σε μια παρεξήγηση που μας κοστίζει 12 εκατομμύρια ευρώ. Απλή ερώτηση ήταν αυτή. Δεύτερη ερώτηση, πιο πρακτική. Ε, τι έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να περιορίσει αυτή τη ζημία. Ποιος ήταν ο υπεύθυνος, τι φταίει δηλαδή, τι διδάγματα μπορεί να εξαγαγεί από την εμπειρία της αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι γίνεται αυτό το καιρό για να αποτραπούν τέτοιες καταστάσεις στο μέλλον. Μου έχουν στείλει πολλές διευκρινήσεις, ορισμένες από τις αμφιβολίες μου διασκεδάστηκαν, αλλά μου γέννησαν καινούριε. Ε, διότι πρώτα απ' όλα η βασική μου αμφιβολία, η βασική μου ερώτηση τώρα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κάτι το οποίο δεν έχω ακόμα ρωτήσει γραπτός γιατί βασίζεται στη νέα πληροφόρηση που μόλις έλαβα. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εάν σε αυτά που λένε εδώ ισχυρίζονται ότι δεν ήταν σαφή ε, ε, η κατάσταση, γιατί λοιπόν δεν κατέθεσε έφεση. Βέβαια, μπορεί να μην είχε τη δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βάλει την απόφαση, αλλά μα το πει για ποιο λόγο δεν το έκανε. Και ένα δεύτερο και πιο σημαντικό ερώτημα. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακόμα και αν είχε αμφιβολίες ή ερωτηματικά, γιατί δεν ακύρωσε το διαγωνισμό όταν είπε η εταιρεία ότι θεωρεί ότι παραβιάζονται τα πνευματικά της δικαιώματα, γιατί δεν ακύρωσε το διαγωνισμό Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, εξ όσων μου απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φαίνεται ότι υπήρξε και διένεξη Έκανε εσωτερική βέβαια αξιολόγηση, ε, ε, έλεγχο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά εγώ ήθελα να μάθω τι πήγε στραβά εκεί για να καταλήξει διαφορετικά το δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Επαναλαμβάνω, το ποσό είναι αρκετά μεγάλο και δεν βλέπω πουθενά έφεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, κανένα από τα στοιχεία που μου διαβίβασαν. Θα με ενδιαφέρει να μάθω βέβαια και τη δική σας άποψη, θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ αγαπητοί συνάδελφοι αν επιτρέπετε, Πρόεδρε, να μας απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν είναι παρόν κανείς από την Επιτροπή να μπορεί να απαντήσει. Θα μας ενδιαφέρει πολύ. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν μπορώ να σας πω όμως ότι είμαι υπέρ μιας τέτοιας μεταφοράς πιστώσεων. Παραμένουν πολλά ερωτήματα ανοιχτά. Euh, Κυρία Συγγετρία, δεν έχουμε χρόνο για ανταλλαγή απόψεων, ούτε καν ανταλλαγή απόψεων με την Κομισιόν. Γιατί έχουμε μια σημαντική συζήτηση για την χρηματοδότηση κτηρίων, πολιτική ακινήτων. Βλέπω ότι έχετε ακόμα ερωτήσεις προς την Κομισιόν. Προτείνω να αναβάλω την απόφαση για την επόμενη φορά. Ο Γενικός Διευθυντής για τις μεταφράσεις της Κομισιόν, ο κύριος Χεργής, δεν είναι παρόν. Δυστυχώ δεν μπορεί να γίνει η συζήτηση σήμερα. Ακούσατε τα ερωτήματα που έθεσε η συγγήτριά μας. Θα μπορούσατε μας τα ήδη από σήμερα το βράδυ διμερός ή γραπτά μέχρι την επόμενη, με το επόμενο ραντεβού να μας δώσετε ικανοποιητικές απαντήσεις έτσι ώστε να συμφωνήσουμε με την μεταφορά που εσείς χρειάζεστε να γίνει. Αυτά ήταν για το 15. 16. Μεταφορές για τα άλλα όργανα. Ελεκτικό συνέδριο. Ράις Δεβρίς, παρόν επιφανές μέλος του Ελληνικού Συνεδρίου. Είχα την ευχαρίστηση και την τιμή να τον γνωρίζω όταν ήταν μέλος του Ευρωκοινοβουλίου πριν από μερικά χρόνια. Μετά επιφανές μέλος της Ολλανδικής Κυβέρνησης, σημαντικός υπουργός στο Συμβούλιο, Έλγα Τρίπελ, η Η πρώτη μεταφορά αγγλικά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αρχίσαμε τη συζήτηση την περασμένη φορά. Εγώ δεν έχω δυσκολίες. Μερικοί συνάδελφοι έθεσαν ερωτήματα και γι' αυτό, μια και είναι παρόν το ελεκτικό συνέδριο, να απαντήσει στις ερωτήσεις αυτές και παρακαλώ τους συναδέλφους να κάνουν ερωτήσεις. Euh, Πρόεδρος, χρόνο για συζήτηση δεν έχουμε. Ράις θα μπορούσατε να, να μας πείτε γιατί είναι σημαντική αυτή η μεταφορά ή ο κύριος Διευθυντής ενδεχομένω. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στο συγγνώμη που δεν να παρόν στην τελευταία συνεδρίασή σας. Αυτή η μεταφορά είναι η εφαρμογή ενός κανονισμού του Συμβουλίου του 77 2 2 90 0 για τις αμοιβέ των μελών του ε, Συμβουλίου, του Ελεκτικού Συνεδρίου και τι γίνεται όταν αντικαθίστανται από νέα μέλη. Είναι μια απλή εφαρμογή αυτού του κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τα ε, οδηπορικά και τα επιδόματα τα οποία πρέπει να πληρωθούν στους, στους, ε, στα μέλη του Ελεκτικού Συνεδρίου όταν αλλάζουν. Η συγγήτρια, τι λέτε, να ψηφίσουμε υπέρ της μεταφοράς. Νομίζω υπήρχε και άλλη μία συνάδελφος που θέλει να ρωτήσει. Η κυρία Βέρτμαν. Ευχαριστώ πολύ. Κατανοούμεν τη βάση αυτής της μεταφοράς πιστώσεων, ωστόσο μου παραμένει αναπάντητο το ερώτημα. Πώς θα μεταφερθεί από εδώ Ε, μάλλον μια μετακόμιση σε μια κοντινή χώρα από εδώ μπορεί να κοστίζει 20.000 ευρώ. Δεν είναι βάση παραστατικών αυτό και αποδείξεων. Είναι κατά αποκοπή. Παίρνεις ένα ε, κονδύλι για τη μετακόμιση. Θα ήθελα περισσότερες προφορίες. Να question, Monsieur Yes, if I can very briefly. εξηγήσω σύντομα Πρώτα πρέπει να έχουμε τα χρήματα στον προπολογισμό, ε, να μπορούμε να τα δώσουμε πριν επιτρέψουμε να γίνουν μετακομίσει. Μετά μιλάμε για μετακομίσει πέντε μελών. Σουηδών και Αυστριακών που θα φύγουν ε, ε, αργότερα μέσα στο 2011 και οι δύο που θα τους αντικαθίσουν. και ο κύριος Ντεβρής, ο οποίος ήρθε στο ελεκτικό συνέδριο στις αρχές του χρόνου. Από κάθε ένα από τα μέλη αυτά έχουμε δύο έως τρεις προσφορές με εκτίμηση τι θα στοιχήσει και πρέπει να έχουμε τα χρήματα στον προπολογισμό. Πρόεδρος, η συγγήτρια τι λέει, τι μας προτείνει. Ίσως δεν χρειάζεται όλο το ποσό και όπως είπα και πριν, η εντύπωσή μου είναι ότι ναι, καλό θα είναι να γίνει αυτή η μεταφορά και εσείς θα σήμερα να ψηφίσουμε υπέρ. Ψηφίζουμε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Τρεις. Αποχές. Μία αποχή αποφασίστηκε μεταφορά. Ικανοποιήθηκε το ελεγκτικό συνέδριο. έργα. ή και μια άλλη μεταφορά για τις υπηρεσίες εξωτερικής δράσης. Αυτό είναι λίγο πιο πολύπλοκο. Και σχετίζεται με το επόμενο σημείο, με τα κτίρια. Γιατί μας ζητάνε για την εξωτερική υπηρεσία να, να προσλάβει άτομα για υπηρεσίες για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης η Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινη Πόρη της Κομισιόν και το Ταμείο του ε, Διατάκτη θα δώσει διοικητικές υπηρεσίες για προσωπικό που θα, θα αποσπαστεί από το Συμβούλιο και νέο προσωπικό και για τα κτίρια θα χρησιμοποιούν επιπλέον προσωπικό σε προετοιμασία για την διαχείριση των νέων κτηρίων της εξωτερικής υπηρεσίας. Τι σημαίνει αυτό. 1,6 εκατομμύρια επιπλέον για την προπαρασκευή της δίκησης για το νέο κτίριο. Ε, για να είμαι ειλικρινής μου φαίνεται λίγο περίεργο αυτό το νούμερο. Οπότε περνάμε και στο επόμενο σημείο, στο σημείο αυτό, τη συζητήσουμε και τα δύο μαζί. Triple. Ναι, ναι, Αν τα πάρουμε μαζί για να έχουμε την πλήρη εικόνα από τους υπεύθυνους. Τι σημαίνει γιατί κατά τη γνώμη μου δεν είναι η πιο σωστή λύση. Και παρά είναι ακριβή. Στο 17 λοιπόν, σε σχέση πάντα με το 16, στρέφουμε στην εισηγήτριά μας, την Μόνικα Ολμάγερ, παρουσία του κυρίου Εύαν, διευθυντής στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης δύο φορές στην Επιτροπή Προπολογισμών. Το συζητήσαμε τώρα πρέπει να πάρουμε θέση. Η κυρία Χολμάγερ. Πρόεδρε, μια και πρόκειται μια πολύ σημαντική απόφαση, επιτρέψτε μου λίγο να εξηγήσω βάσει και των όσων είχαμε συζητήσει ανάμεσα αποφάσεως και πάλι. Πρόκειται για τα, για τα κτίρια Μπρεντέλ 1 και 2 και τη δυνατότητα αντί για ανανέωση της μίσθωσης να διαθέσουμε το ποσό που χρειάζεται για την αγορά του κτίριου. Στο κόστο, στι δαπάνε, αυτά που έχει γράψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είμαι κάπω επιφυλακτική και έτσι δεν θα επισέλθω στα, ποσό, στα ποσά. Δεν θέλω να συζητήσω Άλλωστε δεν είναι και το ουσιαστικό στην υπόθεση αυτή. Σε πέντε περίπου χρόνια το κτίριο αυτό θα χρειαστεί σημαντική ανακαίνιση. Και ασφαλώς τότε θα αυξηθεί και το τίμημα. εκτός του ότι μπορεί να υπάρχουν και επιπλέον μέτρα που θα, θα προκύψουν στην συνέχεια, που θα χρειαστεί να ληφθούν δηλαδή. Ωστόσο έχουμε ω πρόβλημα το χρόνο, δηλαδή μία διαδοχική, μία σειρά, ε, αλλά σειρά μετακομίσεων, φεύγουν κάποιοι άλλοι μπαίνουν κτλ. Και, και έτσι δεδομένου ότι ε, δεν επαρκούν οι χώροι που διαθέτει και το Συμβούλιο, θα πρέπει να προβλεφθεί η μίσθωση νέων κτηρίων. Αυτό ήδη θα σήμαινε και σημαντικές καθυστερήσεις σε με το ΕΑΝΤΕΣ και σημαντικές δυσκολίες. και νομίζω ότι καλό θα ήταν να δούμε τι μπορεί να προκύψει σε περίπτωση που κτίρια που έχουν και ηλικία αρκετών δεκαετιών χρειαστούν ε, κάποια στιγμή απασβέστοση Φερρυπίνη αν προκύψει ότι έχουν ε, απαμιάντωση μάλλον αν ε, αποδειχθεί ότι είναι επιμολυσμένα με αμίαντο και χρειαστεί αυτή η ιστορία και η εξυγίανση των κτίριων. Για τα πραγματικά περιστατικά λοιπόν δεν είναι απλή η απόφαση, αλλά επιλογές δεν έχουμε. Και γι' αυτό διατυπώνω ξεκάθαρα μια θέση και γι' αυτό κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να σημειώσω ότι πρέπει πλέον να μπει ένα τέρμα σε κόλπα τα οποία τελικά μας ξεγελούν, δηλαδή κατατίθενται προτάσεις ε, με το μισό ποσό μόνο στο προσχέδιο του προϋπολογισμού και μόνο όταν επανέλθουμε και ξαναρωτήσουμε και ζητήσουμε διευκρινής για 25η φορά μας δίνουν τα πραγματικά ποσά πράγμα το οποίο είναι ενοχλητικό. Η διερεύνηση δηλαδή των πραγματικών δεδομένων είναι πολύ κουραστική και ενοχλητική, άσχετο των των καλών σχέσεων που μπορεί να έχουμε. Επί παραδείγματι, όταν λέει η Επιτροπή 850.000 τετραγωνικά μέτρα είναι ε, ο χώρος, η επιφάνεια την οποία χρειάζεται και τώρα έχει 18.000 μόνο, τότε δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι μέχρι τα 850.000 τετραγωνικά μένουμε σε ε, πεδίο ουδέτερο δημοσιονομικά. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Ουδέτερος δημοσιονομικά σημαίνει πράγματι δεν προξενείται επίπτωση στον προπολογισμό. Αντικειμενικά και με βάση τα στοιχεία τα ουσιαστικά δεν υπάρχει επίπτωση στον προπολογισμό. Και ως προς την ε, κεφαλαιοποίηση έχουμε εδώ να κάνουμε με μία ε, σύμβαση η οποία δεν είναι ξεκάθαρη, η οποία οδηγεί σε πολλές ανησυχίες και υποψίες 12,5 εκατομμύρια για 25 μήνες χωρίς καταβολή αντιτίμου, μισθώματος δηλαδή. Ωστόσο όμως αυτά τα ποσά δεν έχουν υπολογιστεί πλήρως, διότι δεν έχει υπολογιστεί σε αυτήν την υπόθεση ο εξοπλισμός αυτού του χώρου. Άρα, και δεδομένων των εμπειριών που έχουμε από την Επιτροπή, μπορούμε να, μπορεί να ξεπεράσουμε και τα ποσά αυτά. Ουδέτερα λοιπόν ως προς τον προπολογισμό δεν είναι τα σχέδια αυτά. Ως προς την ασφάλεια επίσης έχουμε ζητήματα και ως προς τον εξοπλισμό των κτηρίων που δεν είναι καθόλου σαφής ακόμη η εικόνα που προκύπτει. Μπορεί να γίνεται λόγος για 20 εκατομμύρια για τον εξοπλισμό και 8,5 για την ασφάλεια. Άρα λοιπόν η απόκληση από κόστο, σημαντική απόκληση από κόστο που έχει προβλεφθεί σε συγκεκριμένε προτάσει, θα πρέπει να ε, προτείνεται με συγκεκριμένη αιτιολόγηση σε κάθε περίπτωση, εφόσον αυτό, όπως είπα, σημαίνει επιβάρυνση με επιπλέον θαπάνες. Ε, εάν όχι, εντάξει, δεν πειράζει, αλλά εάν πρόκειται να αυξηθεί το κόστο, θέλω εξάπαντο να χορηγούνται λεπτομερεί εξηγήσει και αιτιολόγηση. Ω προ την επιφάνεια. 49 49.000 τετραγωνικά, δύο από την Επιτροπή, 12 από το από το Συμβούλιο, 5.000 από την Επιτροπή των Περιφερειών είναι οι επιφάνειες που απελευθερώνονται και η Επιτροπή για το 11, το 12, το 13 έχει ανακοινώσει ότι σκοπεύει να ε, παρετηθεί από την χρήση ορισμένων ε, εγκαταστάσεων, γραφείων δηλαδή, σε ορισμένες περιοχές όπως στην Κόρτενμπερκ 107 και στην Κούχθε Μισελ επίσης. Δεύτερη ερώτηση βέβαια εδώ είναι το τι είδους, ε, τι σημαίνουν ε, συγκεκριμένα αυτά τα ε, γραφεία σε, επιφάνεια συγκεκριμένα και πόσο μπορεί αυτό να είναι ουδέτερο δημοσιονομικά. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται νέες εκτάσεις γραφείων, νέα τετραγωνικά γραφείων, τότε θα πρέπει, και πιστεύω να με υποστηρίξετε κι εσείς, θα πρέπει να με εξηγήσει η Επιτροπή γιατί χρειάζεται πέραν των υφισταμένων τώρα αυτών επιφανειών γραφείων να ε, εξασφαλίσει επιπλέον τετραγωνικά. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε αυτήν την ε, ε, αύξηση της επιφάνειας των γραφείων σε ε, χρήσιμη παρεμπίπτουσα δαπάνη και επίσης θα ήθελα να πω ότι και σε επίπεδο Συμβουλίου έχουμε κατασκευή ενός νέου κτηρίου πολλών χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων έχουμε ένα ποσό, μια, ένα, μια ποσότητα μάλλον τραγωνικών μέτρων που ελευθερώνται σε επίπεδο ε, Επιτροπής των Περιφερειών. Έχουμε το κτίριο Lex και από ό,τι φαίνεται μπροστά μας έχουμε τη μεγαλύτερη επέκταση του χώρου των γραφείων και των εγκαταστάσεων που έχουμε στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ελπίζω το Συμβούλιο να μας υποβάλει μια συγκεκριμένη στρατηγική. Δεν μπορεί συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια να εξαπλώνεται και να μην παρουσιάζει ποτέ μια στρατηγική επιχειρησιακή, ένα επιχειρησιακό σχέδιο. Η Επιτροπή βέβαια έχει υποδειγματική στάση σε αυτό, προσπαθεί πάντοτε να βρίσκει τα φθηνότερα τουλάχιστον κτίρια, έστω και εάν πρέπει να φύγει από το ακριβό ε, την ακριβή γειτονιά των ευρωπαϊκών κτιριών, το Συμβούλιο δεν ακολουθεί την ίδια στάση και πρέπει να πω ότι εγώ προσωπικώς δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει όλοι οι μεταφραστές του να βρίσκονται στο κέντρο των Βρυξελών. Αυτό δεν το έχει, καταλα... δεν το έχει εξηγήσει ικανοποιητικά το Συμβούλιο και γι' αυτό νομίζω ότι θα έπρεπε τα θεσμικά όργανα, είτε πρόκειται για Επιτροπή, είτε για Κοινοβούλιο, είτε για Συμβούλιο, είτε για Επιτροπή των Περιφερειών, να έχουν ένα σχέδιο επιχειρησιακό, ξεκάθαρο, να μας ε, υποβάλουν έτσι ώστε να έχουμε μια σεφέστερη εικόνα και επισκόπηση της στρατηγικής και της πολιτικής για τα κτίρια. Κλείνω, Πρόεδρε. Ξέρω ότι προσελκύω πάνω μου τα πειρά των συναδέλφων όταν είμαι τόσο σαφής, αν και ακόμα και αν δεν είμαι τόσο σαφής πάλι δεν τη λιτώνω. Εγώ προτείνω λοιπόν τη λύση παριθμών 1, αλλά παρακαλώ την Επιτροπή μας ιδιαίτερα, ιδιαίτερα ε, επιμένω να μιλήσουμε ναι υπέρ το, του κεφαλαίου των κτηρίων, αλλά να θέσουμε τους δικούς μας όρους. Εάν αναβληθεί η επέκταση του ε, άντες ε, καθυστερεί για αρκετούς μήνες και νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να είναι κάτι επιθυμητό, δεδομένου ότι έχει ξεκινήσει με πολύ κακούς ιόνους του ΕΑΝΤΕΣ ούτως ή άλλως. Ας ελπίσουμε ότι θα βελτιωθεί το κτίριο σε σχέση με αυτά που βλέπουμε τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία εισηγήτρια. Ε, σας ζητώ συγγνώμη για λόγους ε, ε, χρονικού Ο κύριος Μάνκα έχει το λόγο. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. η κυρία Χολμάγερ έκανε μια έκθεση ε, έχει κάνει πολύ σωστά συμπεράσματα από τα στοιχεία που είχε όμως στα χέρια της. Αν δούμε όλα τα στοιχεία ε, θα καταλάβουμε ότι αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστός τρόπος λειτουργίας. Δεν έχουμε ε, όλα τα στοιχεία για τη διαπραγμάτευση, ε, δεν έχουμε τις αναλεκτικές προτάσεις στα χέρια μας, μόνο το μίσθωμα και την αξία. Αλλά αν δεν έχει κάποιος εναλλακτικές ε, προτάσεις, δεν έχει και περιθώριο ελιγμών. Και αν δεν το δημιουργεί, δεν είναι επαγγελματία. Αυτή τη φο... Ε, πρέπει να σας πω ότι όταν κάποιος δεν έχει τα προσόντα και τις δυνατότητες, πρέπει να ασχολείται με κάτι άλλο, να μην προκαλεί ζημίες. Όταν εγώ δεν είχα εναλλακτική λύση απέναντι στην κοινή γνώμη, τη δημιούργησα και άρχισα να με σέβονται ως συνομιλητή. Ε, επίσης είμαστε σε μια κατάσταση που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας την καλή βούληση και του ιδιοκτήτη, αλλιώς θα έχουμε πολλά προβλήματα και οικονομικά και άλλα. Εγώ δεν έχω άλλη λύση παρά να υποστηρίξω και την εισηγήτρια και την ε, πρόταση αυτή και τη γνωμοδότηση, ε, αλλά θα πρέπει να κάνουμε και κάτι άλλο ως πρόταση, να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να δεσμευτεί όμως και το Κοινοβούλιο ότι στο μέλλον δεν πρόκειται να κάνει τέτοιες ε, ενέργειες. Ο κύριος Χάρτονγκ, μία φράση μόνο. Πρόεδρε, μία φράση. Εγώ δεν επιλέγω ούτε την επιλογή 1 ούτε την επιλογή 2. Παρακαλώ να σημειωθεί ότι καταψηφίζω ολόκληρη ε, την πρόταση διότι θα σημαίνει τεράστια αύξηση του κόστου. Ευχαριστώ πολύ. Λογικό. Η κυρία ε, Φέρτμαν, ναι ή όχι. Äh, ε, θα ήθελα παρόλα αυτά να τονίσω ότι δεν έχουμε δετερότητα ως προς το κόστος όπως μας είχαν υποσχεθεί ε, τιμή εξαγοράς που είχαμε βάλει ως στόχο δεν επετεύθη, ούτε ένα δευτερόλεπτο δεν το συζήτησαν μαζί μας και έχουμε πολύ μεγάλες δυσκολίες να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Τα συζητήσαμε όλα αυτά πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Το τελευταίο σημείο που έπρεπε να διευκρινιστεί είναι αν μπορούμε να παίξουμε το χαρτί της Μπελιάρ. Ε, Μπρεντέλ, διορθώνει ο Πρόεδρος, όχι Μπελιάρ. Ε, η συγγήτρια μας λέει όχι γιατί ε, σημαίνει επιπλέον κόστος και επιπλέον χρόνο. Ε, το έχουμε εξαντλήσει το θέμα. Ο κύριος Άγγλων θα μας πει ναι ή όχι η κυρία Γκρέσλε και μετά να ψηφίσουμε παρακαλώ. Έγκλοντ, ε, πρόεδρε, ε, πώς καταλήξαμε πάλι σε αυτή την κατάσταση που πιεζόμαστε να αποφασίσουμε για λόγους χρονικούς. Είναι παράλογο αυτά τα πράγματα. όλοι δυσκολευόμαστε. Ναι, ο πρόεδρος. Σε ένα λεπτό θα φύγουν οι διερμηνείς. Ναι, ναι, εντάξει, καλά, καλά. Και αυτό παράλογο είναι. Ότι συζητάμε ένα τόσο σημαντικό θέμα και πρέπει να τελειώσει η συνεδρίαση. Εγώ δεν μπορώ να σας πω. Ε, δεν, θέλω να πω δέκα πράγματα. Εάν δεν μπορούμε να τα πούμε, δεν μπορώ να ε, πάρω απόφαση και δεν μπορώ να το υιοθετήσω. Ο πρόεδρος. Όσου διαμαρτύρεστε ότι δεν είχαμε χρόνο, σα θυμίζω ότι έχουμε εξαντλήσει και υπερβεί κατά πολύ τι προθεσμίε που προβλέπει ο κανονισμό του Κοινοβουλίου για να γνωμοδοτήσουμε. Το έχουμε εξαντλήσει το θέμα. Αυτό που σήμερα συζητούμε είναι απλώ η επιλογή Μπραντέλ. Ε, κάποια στιγμή για ένα θέμα τόσο σημαντικό θα πρέπει η Επιτροπή Προπολογισμών να μπορεί να είναι σε θέση να λάβει απόφαση. Η κυρία Ντουρόν. Θέλω να πω μόνο ότι μα ζητούν σήμερα να επιλέξουμε ανάμεσα στην πανόλη και τη χολέρα, μπρο γκρεμό και πίσω ρέμα. Δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα. Και παρακαλώ την επόμενη φορά να έχουμε ένα πλάνο, ένα σχέδιο. Εγώ είμαι μέλος του Προεδρείου ε, του Κοινοβουλίου για τα κτίρια. Ε, κάθε φορά μας ζητούν ε, να λογοδοτούμε και το κάνουμε. Παρακαλώ το ίδιο να κάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Γκρέσλε. Μα εμείς δεν ξέρουμε αν ε, ενδείκνυται το κτίριο αυτό, το κάπιτα. Και ποιο είναι το επιπλέον κόστος, ποια είναι τα εμβαδά, ποιο είναι το, το δυναμικό. Αν δεν τα έχω όλα αυτά τα στοιχεία στα χέρια μου δεν μπορώ να υπερψηφίσω. Ο πρόεδρος. Κοιτάξτε αγαπητοί συνάδελφοι. Μήνες ολόκληρους όλες οι πολιτικές ομάδες κατηγορούν την κυρία Άστον και την υπηρεσία της για αδράνεια, για αναποτελεσματικότητα ε, και ε, για αβελτηρία. Ε, αυτό το έχουμε συζητήσει τόσο πολύ καιρό. Δεν έχουν λυθεί τα πάντα. Αν είχαμε όσο χρόνο θέλαμε στη διάθεσή μας θα μπορούσαμε να τα έχουμε λύσει όλα αυτά. Δυστυχώς έρχεται η στιγμή να αποφασίσει κανείς μια ώρα. Τώρα... Εισηγήτρια, ποια, τι συνιστά. Εγώ είμαι υπέρ της επιλογής υπαριθμών 1 ε, με την επιφύλαξη όλων αυτών που σας κατέθεσα. Και θα παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών να δεσμευτούν ότι θα τα τηρήσουν. Και αγαπητοί συνάδελφοι κυρία Γκρέσλε, δεν χρειάζεται το κτίριο Capital. Το έχω επισκεφθεί στο μεταξύ δεν είναι απαραίτητο. Το κτίριο Μπρεντέλ έχει και αυτό προβλήματα ασφαλείας. Είναι δίπλα ε, σε ένα βενζινάδικο. Τώρα δεν ξέρω ε, ε, είναι το ίδιο με το σούπερ μάρκετ. Τι να κάνω, εγώ μπορώ να επιλέξω μεταξύ των επιλογών που μου δίνουν και τίποτα παραπάνω. Και αυτό που εκφράζω δεν είναι επιθυμία, είναι απέτηση για ένα μακροχρόνιο πολιετή σχεδιασμό όχι μόνο του Κοινοβουλίου αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Επιτροπής Περιφερειών. Γιατί αυτά τα πράγματα εδώ είναι εκτρά ως διαδικασίες. Ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, θέτω την πρόταση της ηγήτριάς μας ποιος είναι υπέρ της επιλογής υπαριθμών 1. 16. Qui est contre 16. Κατά. Επτά αποχές. Τέσσερις. Ε, ευνοϊκή λοιπόν γνώμη ε, με την πρώτη πρόταση. Τελευταία. Κυρία εισηγήτρια, πιστεύετε ότι για την πίστοση μπορούμε να αποφασίσουμε τώρα ή χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Υποθέτω χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Ωραία. Α, θα ψηφίσουμε την άλλη φορά. Συγγνώμη που σας πίεσα λίγο, αλλά έπρεπε οπωσδήποτε να αποφασίσουμε σήμερα. Ο κύριος Οσάλιβαν δεν ε, πήρε το λόγο, αλλά πήρε τα χρήματα. Λήξη συνεδρίαση, παρακαλώ να παραμείνουν οι συντονιστές.